Bonjour. Καλημέρα σας. Ξεκινούμε την ε, συνεδρίασή μας. Παρακαλώ καθίστε. Έχουμε τη χαρά σήμερα το πρωί να έχουμε μαζί μας την κυρία Ηλιάνα Ιβάνοβα, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Από το 2016 είστε η πρόεδρος του δεύτερου τμήματος, τμήμα το οποίο έχει επιφορτιστεί με το καθήκον του ελέγχου των δαπανών στις διαρθρωτικές δαπάνες, στην ενέργεια και στις μεταφορές. Είναι ένα πολύ σημαντικό θεσμικό όργανο το ελεγκτικό συνέδριο για την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι εκθέσεις που συντάσσει είναι πάντοτε εξαιρετικά διαφωτιστικές και καλύπτουν πεδία τα οποία δεν είμαστε εμείς σε θέση στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή να καλύψουμε. Μετά τη δημοσίευση της έκθεσής σας για τη δημοσιονομική χρήση 2018, θέλησα πολύ γρήγορα να σας καλέσω και να προβούμε σε μια ανταλλαγή απόψεων για να παρουσιάσετε στα μέλη της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής τις εργασίες του δικού σας θεσμικού οργάνου καθώς και τα βασικά συμπεράσματα και συστάσεις. Επίσης θεώρησα ότι θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή σας για τις πρόσφατες εκθέσεις που έχει δημοσιεύσει το ελεγκτικό συνέδριο για την υλοποίηση, την εφαρμογή και τις επιδόσεις και τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής. Χθες στη συνάντηση που είχαμε μιλήσαμε για τα ποσοστά σφάλματος ή τις συχνότητες σφάλματος. Όλα αυτά έχουν βελτιωθεί και μάλιστα κατά πολύ. Παρόλο που ε, παραμένουν πράγματα που πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε ε, σε μια άρτια κατάσταση. Βεβαίως, πάντοτε πρέπει κανείς να έχει υπόψη του ότι η ουσία θα πρέπει να είναι απλουστευμένη για τους δικαιούχους και είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία σε αυτή τη λογική της ε, ε, διαμοιρασμένης διαχείρισης. Είναι μεγάλη χαρά για μας που θα σας ακούσουμε να παρουσιάζετε το σύνολο αυτών που κάνετε και το σύνολο των συστάσεων. Βεβαίω αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για εσά, γιατί δεν θα έχετε αρκετό χρόνο στη διάθεσή σα. Σα διαβεβαιώ όμω ότι αυτή η συζήτηση είναι η πρώτη από μια σειρά συναντήσεων που θα έχουμε μαζί εσεί και εμεί καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη κοινοβουλευτική θητείας και έχουμε την πρόθεση ε, να κάνουμε το παν για να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του Ελεκτικού Συνεδρίου και τη δική μα κοινοβουλευτική επιτροπή για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τι Περιφέρειε. Θέλω επίση να υπογραμμίσω δημόσια την εξαιρετική συνεργασία του διοικητικού προσωπικού της Επιτροπής μας με τους ομολόγους τους, το αντίστοιχο διοικητικό προσωπικό του ελεγκτικού συνεδρίου. Είπατε ότι το ποσοστό σφάλματος πέρασε από το 3% στο 5% από το 15-17 μέχρι και το 18%. Όμως πριν το 2015 ξεπερνούσε το 10%. Άρα η ανάλυση σας για τα μέλη της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής θα είναι εξαιρετικά εμπεριστατωμένη. Ε, θα την λάβουμε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη γιατί την ε, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική. Και πρέπει να μιλήσουμε και για κάποια στερεότυπα που βαραίνουν την πολιτική συνοχή και νομίζω ότι οι αριθμοί θα τα διαψεύσουν. Έχω την εντύπωση ότι επιδιώκοντας δίκαιους σκοπούς για, για να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που έλεγε χθες ο συνάδελφος Νοβάκοφ, να ε, εξαλείψουμε τα λάθη, έτσι θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την πολιτική συνοχή. Έχετε το λόγο για 20 λεπτά κυρία Ιβάνοβα και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να γίνει συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ μεγάλη χαρά να είμαι εδώ στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για να παρουσιάσω τη δουλειά μας στο αντίστοιχο αρμόδιο τμήμα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πράγματι σας ευγνωμονώ ε, θα περάσω στα αγγλικά. Πριν ξεκινήσω, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για αυτούς που ήδη γνωρίζουν αυτά τα θέματα. Ίσως θα κουραστούν και θα θεωρήσω ότι είναι ε, επαναληπτικά. Θα κάνω το πάνω όμως μέσα στα 20 λεπτά να ε, μιλήσω για τη συμμόρφωση για την νομοτήτα, για την νομοτυπία των ευρωπαϊκών δαπανών. Στη συνέχεια θα μιλήσω για τις επιδόσεις, για ε, τις διάφορες ειδικέ εκθέσεις που συντάσσουμε και εκπονούμε στο ελεγκτικό συνέδριο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω καταρχάς δύο λόγια για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε οργανωθεί. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει αναθέσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου του σε πέντε τμήματα. Κάθε τμήμα αποτελείται περίπου από πέντε μέλη και έχει επιφορτιστεί με το καθήκον να μελετά συγκεκριμένο κλάδο ευρωπαϊκών δαπανών, συγκεκριμένο τομέα. Εγώ είμαι υπεύθυνη για τη μελέτη των δαπανών για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και απασχόλησης Συχνά αναφέρεται αυτό ως συνοχή. Υπάρχει το τμήμα 1 για τη γεωργία, το τμήμα 3 για τις δαπάνες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί καλύπτουν διάφορους τομείς πολιτικής και βλέπετε ότι εμείς καλύπτουμε τρία από τα ε, πέντε ευρωπαϊκά ταμεία, διαθροτικά και επενδύσεων και συνοχής. Πολλά, πάρα πολλές οι δαπάνες είναι ε, αυτές που εντάσσονται στο δικό μου αρμόδιο τμήμα. Κάνουμε δύο είδη ελέγχων στο ελεγκτικό συνέδριο. Έλεγχο συμμόρφωσης, πρώτον, compliance audit. Ελέγχουμε κατά πόσο οι ευρωπαϊκές δαπάνες ε, ε, ευθυγραμματίζονται με τους συγκεκριμένους κανόνες, ο έλεγχος επιδόσεων, performance audit, ξεπερνά όλο αυτό. Δηλαδή βλέπουμε κατά πόσο οι δαπάνες ε, έδωσαν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, κατά πόσο έγιναν με εύλογο κόστος, λογικό και κατά πόσο πράγματι βελτίωσαν τη ζωή του Ευρωπαίου πολίτη. Επίσης ε, δημοσιεύουμε γνωμοδοτήσεις για προτινόμενη νομοθεσία, δημοσιεύουμε ανακοινώσει και αξιολογήσεις που δεν περιλαμβάνουν έλεγχο αυτό καθεαυτό αυτό, αλλά εκτιμήσεις και αναλύσεις. Και θα μιλήσω στη συνέχεια για αυτά τα παραγόμενα ε, προϊόντα του ελεγκτικού συνεδρίου. Ας δούμε τους ελέγχους συμμόρφωσης. Κύριε Πρόεδρε, στην ετήσια έκθεση το είπατε κι εσείς, ε, δημοσιεύονται ετησίω τα αποτελέσματα των ελέγχων μας, είναι ετήσια η χρήση, άρα τα αποτελέσματα για τα 2019 δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα είναι η δήλωση ε, βεβαιότητας διασφάλισης, Statement of Assurance, το περιβόητο DAS. Και μιλούμε για την ομοτυπία και την ομότητα των δαπανών στη συνοχή. Έχουμε ένα μέλος που κάνει αυτές τις εκθέσεις, ο Τόνι Μέρφυ, ο Ιρλανδός συνάδελφος, ο οποίος θα παρουσιάσει τα ευρήματα του έκτου κεφαλαίου στην αντίστοιχη Επιτροπή ΚΟΡ την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, εγώ θα κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις σήμερα, γιατί την επόμενη εβδομάδα ο Ιρλανδός συνάδελφος θα κάνει λεπτομερή παρουσίαση επί της ουσίας της έκθεσης. Από τις διαφάνειες όμως βλέπετε και παρατηρείτε ότι το επίπεδο σφάλματος, η αναλογία δαπανών που δεν συμμορφούνται με τους κανόνες, ήταν στο 5% του 2019 είναι το επίπεδο αυτό σφάλματο ψηλότερο από το συνολικό επίπεδο σφάλματων σε σχέση με τον ευρωπαϊκό Προπολογισμό και ψηλότερο σε σχέση με την περσινή χρονιά, πολύ σωστά τα είπατε κύριε Πρόεδρε. Ποιο είναι ο βασικός λόγος. Το γεγονός ότι οι δικαιούχοι στα κράτη-μέλη ζήτησαν project μη επιλέξιμα, οι δαπάνες μη επιλέξιμες και Νομίζουμε ένα από τα πράγματα που θα μπορούσε να βοηθήσει για να μειωθεί το επίπεδο σφάλματος και το διοικητικό άχθος είναι η απλούστευση ορισμένων των, από τους κανόνες. Και θα ήθελα σε αυτό το στάδιο να αναφερθώ και να πω ότι εμείς στο τμήμα 2 πιλωτικά υλοποιούμε μια νέα προσέγγιση σε σχέση με τους ελέγχους συμμόρφωσης τα τελευταία δύο χρόνια και την λέμε έλεγχο βεβαίωσης, attestation, πιστοποίησης αν θέλετε. Δηλαδή προσπαθούμε να βεβαιώσουμε καλύτερα το έργο άλλων οργανώσεων σε σχέση με τις διαδικασίες ταπανών και στα κράτη-μέλη και εντό Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Είναι πολύ τεχνικό αυτό το ζήτημα και δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα περιοριστώ αυτά στο, σε αυτά για το, ε, την ετήσια έκθεση και το τμήμα 6. Απλά ένα στιγμιότυπο σας παρουσιάζω αυτή τη νέα προσέγγιση με τη βεβαίωση, attestation. Γιατί βλέπουμε αυτούς τους χάρτες τώρα, για να δείτε το, το έργο, το φόρτο εργασίας μας καλύπτουμε δύο περιόδους δαπανών, 2007-2013 και 2014-2020. Βεβαίως είναι πολλές οι πληροφορίες. Το βασικό όμως είναι ότι οι 220 ατομικές συναλλαγές που εξετάστηκαν προέρχονται από διαφορετικά κράτη-μέλη και ήταν απαραίτητες και εξαρτάται από την ποιότητα της δουλειάς που έγινε από τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη. Σε κάθε περίπτωση εμείς παρακολουθούμε την πορεία του ευρωπαϊκού χρήματος μέχρι και τον τελευταίο τελικό αποδέκτη. Προσοχή όμως. Ο έλεγχος συμμόρφωσης έχει σχεδιαστεί για να παρέσχει συμπεράσματα για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, για τον τομέα πολιτικής. Δεν θα δείτε το ατομικό επίπεδο σφάλματος ανακράτος μέλος. Ξέρω ότι το θέμα αυτό σας ενδιαφέρει και πολύ συχνά μας θέτετε ερώτηση για τη χύψη χώρα, αλλά εμείς δεν είμαστε σε θέση να εξάγουμε συμπεράσματα για τα ατομικά επίπεδα σφάλματος για το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Πρέπει να γίνει πολύ περισσότερη δουλειά για να υπάρξουν στατιστικώς χρήσιμες και αξιόπιστες ε, εκτιμήσεις και συμπεράσματα για τα επίπεδα ασφάλματος ξεχωριστά ανά συγκεκριμένο κράτος μέλος. Στρέφουμε τώρα στο τομέα των επιδόσεων, έλεγχος επιδόσεων, performance audit. Εδώ διαλέγουμε τα αντικείμενα του ελέγχου μας. Εκεί πιστεύουμε ότι τα διαλέγουμε με βάση τα κριτήρια που πιστεύουμε ότι θα μας φέρουν μεγαλύτερη αξιοπιστία και μεγαλύτερη χρησιμότητα. Βλέπετε κάποια, κάποιους τομείς που έχουμε διαλέξει, μια καλή ποικιλία θεμάτων. Έχουμε τα ΣΔΙΤ, έχουμε τις ευρυζωνικές συνδέσεις, έχουμε την ε, απορρόφηση της νομοθεσίας, την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, το ποσοστό απορρόφησης, ε, του σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας, τα δικαιώματα των επιβατών, την απάτη, την ηλιακή και αιωλική ενέργεια. Προσωπικά επί... βλέπω έναν έλεγχο για την αστική κινητικότητα που θα δημοσιευθεί του χρόνου. Και παρόλο που πολλά χρήματα δίδονται για αυτά τα σημαντικά ζητήματα, εναπόκειται στις πόλεις, στους δήμους να τα αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Άρα έχουμε διαχείριση έργου την οποία μοιραζόμαστε και πολύ μεγαλύτερες και περισσότερες προκλήσεις από ότι όταν έχουμε να κάνουμε με οριζόντια προγράμματα, ειδικά από πλευράς επιδόσεων. Εδώ αναφέρω μία από τις προκλήσεις που έχουμε, τον στόχο των 13 μηνών. Τι είναι αυτό. Ε, πιέζει ο χρόνος. Η συμμόρφωση που εξετάζουμε σε σχέση με τις εκθέσεις μας που αφορούν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βάσει χρηματοπιστωτικού κανονισμού και χρηματοοικονομικού και έχουμε ένα μέγιστο όριο 13 μηνών με βάση τον κανονισμό και αυτό είναι τεράστια πρόκληση για μας, για ένα τμήμα σαν και το δικό μας όπου ε, η διαχείριση είναι διαμοιρασμένη, τη μοιραζόμαστε ε, εργαζόμαστε σε επίπεδο κράτους μέλους. Μπορούμε να διαλέξουμε να μην επισκεφθούμε ένα κράτος μέλος όμως αν δεν επισκεπτόμασταν ένα κράτος μέλος οι εκθέσεις μας θα ήταν πολύ λιγότερο ενδιαφέρουσες και πολύ λιγότερο εκτεταμένες. Άρα χρειάζεται αρκετός χρόνος για να ολοκληρωθούν και να γίνουν όλα αυτά. Εργαζόμαστε σκληρά για να ανταποκριθούμε σε αυτό το στόχο και σε αυτή την πρόκληση. Δεν είναι όλα τα προϊόντα που παράγουμε εκθέσεις ελέγχου. Εκδίδουμε και γνωμοδοτήσεις και αναθεωρήσεις και ενημερωτικά σημειώματα όταν μας το ζητούν. Υπάρχει ένας μηχανισμός που ακολουθούμε που προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οι νομοθετικές αρχές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να ζητήσουν τη γνώμη μας για συγκεκριμένη νομοθεσία που μπορεί να έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εμείς συντάσσουμε έκθεση ή γνωμοδότηση. Ένα παράδειγμα πέρσι η γνωμοδότηση για το Common Provisions Regulation, για τον ε, κανονισμό κοινών ε, διατάξεων που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ε, ήμουν προϊσταμένη, ε, επέβλεψα προσωπικά την εκπόνηση της γνωμοδότησής μας για τα θέματα αυτά και θα σας πω και περισσότερα λόγια στη συνέχεια για αυτό το θέμα. Τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε να εκδίδουμε προϊόντα επισκοπήσεων ε, με διάφορα αντικείμενα και δεν ε, περιλαμβάνουν ε, κλησεις δεν είναι εκθέσεις ελέγχου. Όποιος και αν είναι ο σχετικός ορισμός, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις ή αποφάσεις αλλά παρουσιάζουν πληροφορίες ε, για συγκεκριμένα θέματα με έναν ε, προσβάσιμο τρόπο για τα ενδιαφερόμενα μέρη και πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμα κυρίως ε, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, όταν δηλαδή προσπαθούν να βοηθήσουν τους νομοθέτες να λάβουν τη σωστή απόφαση. Παραδείγματα επισκοπήσεων φετινών εξετάζουν το πώς δίνονται οι πόροι από τα ταμεία συνοχή ε, στα κράτη-μέλη. Δηλαδή, ε, μιλάμε ε, και για μία μελέτη που δημοσιεύτηκε νωρίτερα φέτος και στο βαθμό που ο βαθμός του σχεδιασμού και της εκτέλεσης επικεντρώνεται στις επιδόσεις. Εδώ θα πω δύο λόγια σε λίγο. Αν ξεκινήσουμε τώρα με τη γνωμοδότηση που σας είπα είναι κάπως παλιά αλλά κάλυπτε ε, σε μεγάλο βαθμό το νομοσχέδιο και μια σειρά κανόνων που θα ίσχυαν σε μια σειρά διαρθρωτικών ταμείων και φυσικά η ίδια γνωμοδότηση επίσης ε, ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και τεχνική αλλά φυσικά αν ενδιαφέρεστε σας συστήνω να τη διαβάσετε. Έχουμε κάποια συμπεράσματα για κάποια κύρια στοιχεία αυτού του νομοσχεδίου. Ξεκινάμε με την απλούστευση. Εδώ, όπως σας είπα, συμπεράναμε ότι γενικά είναι κάτι καλό, αλλά η απλούστευση των κανόνων μπορεί να παρουσιάσει και κινδύνους σε ό,τι αφορά και τη συμμόρφωση αλλά και την εύρωστη οικονομική διαχείριση και αναφέρομαι στις επιδόσεις. Πρέπει να βρούμε την ορθή ισορροπία λοιπόν μεταξύ της απλούστευσης και της διατήρησης του ελέγχου που είναι σημαντικός για το θέμα των επιδάσεων. Επίσης, ε, είναι σημαντική και η ευελιξία στον επταετή προϋπολογισμό η Κομισιόν ε, είχε προτείνει ένα πρόγραμμα σε δύο στάδια και αυτό αυξάνει την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο να απαντήσει στις ε, αλλαγές, όμως χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις σε κάποια project και ανησυχούμε για το επίπεδο της διοίκησης. Το επόμενο πολύ σημαντικό σημείο που συζητήσαμε και χθε ήταν η ευθυγράμμιση μεταξύ τη ε, Ευρωπαϊκής χρηματοδότηση και των Ευρωπαϊκών Προτεραιοτήτων. Αυτό το έχουμε σχολιάσει πολλάκι. Και ενώ έχουν γίνει κάποια βήματα, ένα ισχυρότερο δεσμό μεταξύ τη ε, χρήση τη χρηματοδότηση και του Ευρωπαϊκού Ξαμήνου, πιστεύουμε και ιδίως ε, εφόσον απουσιάζει μία στρατηγική υψηλού επίπεδου για να επιτευχθεί η στρατηγική του 2020 είναι πολύ μεγάλη παράληψη. Ίσως να υπάρξει αυτή η στρατηγική. Στο μέλλον όμως θα έχει αποφασιστεί η χρηματοδότηση. Και εδώ έχουμε σοβαρές ανησυχίες. Και τέλος για τη λογοδοσία, να πω δύο λόγια. Η πρόταση την να ε, ε δώσει αυτή την ευθύνη περισσότερο στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή και να μειώσει τον ε, ρόλο της Κομισιόν και εδώ βλέπουμε ότι κάποιες αντιζηθετήσεις μπορεί να ε, σημαίνουν αυξημένου κινδύνους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ε, σας είπα, είναι αρκετά μακροσκελής η γνωμοδότηση και τεχνική, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Τώρα, να περάσω σε ένα από τα προϊόντα της επισκόπησης, όπως σας είπα και νωρίτερα. Πρόκειται για την κατανομή των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής 2021-2027. Μην σοκαριστείτε από αυτή την εικόνα, δεν ε, πρόκειται τώρα να σας την εξηγήσω για να την ε, καταλάβετε, αλλά απλώς θέλω να σας δείξω την πολυπλοκότητα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία και ο στόχος αυτής ε, της επισκόπησης ήταν να βοηθήσουμε τα ενδιαφερόμενα μέλη να καταλάβουν τη λογική πίσω από τις διαδικασίες, πώς λειτουργούν δηλαδή. Φυσικά αναγνωρίζουμε ότι η Κομισιόν ήταν πολύ πιο διαφανής σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Δημοσιεύει τις προτάσεις στον κανονισμό CPR που σας ανέφερα νωρίτερα, κανονισμό περί κοινών διατάξεων, όμως είναι πολύ δύσκολο, ακόμη και για μας και για μένα, να καταλάβω, δηλαδή ήταν πρόκληση να καταλάβω τη διαδικασία και κατόπιν να τη μεταφράσω με έναν κατανοητό τρόπο και να την εξηγήσω. Ελπίζουμε ότι αυτή η επισκόπηση δεν είναι τόσο μακροσκελής όπως για το CPR, είναι ένα πιο συντομόγραφο, αλλά θα βοηθήσει τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή τους νομοθέτες και ιδίως το Κοινοβούλιο να λάβει πιο ενημερωμένες αποφάσεις. Εδώ Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των προτάσεων της Κομισιόν στα διάφορα Δεν πρόκειται για νέες πληροφορίες. Μια απεικόνηση απλώς έχετε εδώ. Έχουμε κάποια νέα στοιχεία στη νέα πρόταση. Έχουμε ενότητα όρια ε, και ασφαλείας ε, όπου έχουμε περιορισμούς για την επόμενη περίοδο. Έχουμε έξι κρατή-μέλη που βάσει της πρότασης θα λάβουν τα ίδια ποσά χρηματοδότησης για την πολιτική συνοχή. Υπάρχουν και κάποιες σημαντικές ε, τροποποιήσεις για άλλα κράτη-μέλη, έχουμε νέα στοιχεία όπως μετανάστευση, κλιματική αλλαγή, Έχουμε νέα στοιχεία και βελτίωσεις, όπως σας είπα. Ε, το συμπέρασμα είναι ότι εξακολουθούν να είναι πολύπλοκα τα πράγματα και μπορεί να δοθεί η εντύπωση ότι δεν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Υπάρχει όμως βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους. Τώρα στη δεύτερη ε, σκόπιση που είναι πιο καινούρια και την δημοσίευσαμε πιο πρόσφατα εξετάζουμε σε ποιο βαθμό η πολιτική συνοχή αντικατοπτρίζει τις επιδόσεις και όχι μόνο τη συμμόρφωση. Η κύρια βάση για το έργο μας εδώ ήταν ε, μια δική, όλες μάλλον οι ειδικέ εκθέσεις, 69 εκθέσεις συνολικά που δημιουργήσαν τα τελευταία έτη σε διάφορους τομείς πολιτικής, από τις μεταφορές μέχρι την κοινωνική πολιτική, τις υποδομές, πάρα πολλές εκθέσεις. Και για να διαθρώσουμε αυτό το έργο έχουμε χωρίσει σε πέντε στάδια τον κύκλο της εφαρμογής από το στρατηγικό σχεδιασμό μέχρι την αξιολόγηση. Κατόπιν εντοπίσαμε 14 κατευθυντήριες γραμμές που πιστεύουμε είναι βασικές έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση εξυπηρετεί τις επιδόσεις. Οι 13 ε, καλύπτουν τα 5 στάδια και ο τελευταία κατευθυντήρια γραμμή είναι πιο οριζόντια, βιωσιμότητα και φυσικά είναι οριζόντια για τις φύσεις της. Στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε ότι χρησιμοποιήσαμε τα χρώματα του φαναριού, ε, του, του φωτεινού σηματοδότη. Μπορείτε να δείτε εδώ ε, πιο εύκολα τη σύγκριση μεταξύ των ε, περιόδων και φυσικά εδώ έχουμε και την περίοδο 2021-2027 που είναι ακόμα στο σχεδιασμό και συγκρίναμε το βαθμό στον οποίο οι αρχές αυτές γίνονται σεβαστές. βλέπετε βάσει χρωμάτων ότι υπάρχει σαφής βελτίωση μεταξύ πρώτης και τελευταίας περίοδου. Έχουμε περισσότερα κόκκινα στην πρώτη περίοδο που τώρα έχουν εξαφανιστεί, αλλά βλέπετε ότι οι βελτιώσεις ε, γίναν ε, μεταξύ του 2007 και του 2014 και δεν υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση μεταξύ δεύτερης και τρίτης στήλης. Και αυτό συνάδει με την γνωμοδότησή μας ε, για το CPR που σας ανέφερα πριν δεν περιοριζόταν ε, σε πτυχές επιδόσεων, αλλά το συνολικό μήνυμα ήταν παρόμοιο ότι μπορεί να μην συνεχίζεται αυτή η ορμή που είχαμε για βελτίωση προς την επόμενη περίοδο. Ελπίζω να κάνω λάθος. Όμως τα συμπεράσματά μας ε, είναι αυτά που βασίζονται στις 69 ειδικέ εκθέσεις, όπως σας είπα, της τελευταίας δεκαετίας. Και οι δύο αρχές που αξιολογήσαμε ε, για την περίοδο 2021-2027 θα σας αναφέρω είναι σημαντικές, έχουμε σημαντικές βελτιώσεις, είναι σαφές, τις αναγνωρίζουμε, τις εκτιμούμε, αλλά αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά στοιχεία και η υπαριθμόν ένα κατευθύνια γραμμή είναι το πιο σημαντικό μήνυμα. Αφορά την ανάγκη για στρατηγικό όραμα για την καθοδήγηση των δαπανών. Όταν ε, νωρίτερα αναφέρθηκα στην κομμαδοτησή μα για το CPR, είπα ότι τονίσαμε ότι υπάρχει ε, μία απουσία, δεν υπάρχει διάδοχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι είχαμε υπαναχωρήσει από αυτή την αρχή, από το κίτρινο στο κόκκινο. Επίσης, ε, σημειώσαμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να εργάζεται σε μια σειρά διάφορων στόχων που μερικές φορές είναι ανταγωνιστικοί και δεν είναι ευθυγραμμισμένοι μεταξύ τους. Ε, μιλάμε και για το είναι επτάτη περίοδο του πολιτικού δημοσιονομικού υπηρεσίου, επίσης το σχέδιο Juncker, τις εξωτερικές αναλήψεις υποχρεώσεων, όπως το έχει βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλούς στόχους εδώ και εκεί, όμως ε, δεν υπάρχει μια συνεκτική στρατηγική, ένα συγκεκριμένο όραμα με μετρήσιμους στόχους για το μέλλον, προς το παρόν. Και η κατευθύρια γραμμή 9 αφορά την αναθεώρηση των προγραμμάτων. Ο κίνδυνος εδώ είναι ότι μπορεί να θεωρηθούν τα προγράμματα των κρατών μελών χωρίς ε, να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της επιδόσης. Το νομοθετικό πλαίσιο ενδυναμώθηκε ε, μέσω της αγωγής ε, της ανάγκης για να μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μαζί με τους κανόνες στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 και για το 2021-2027 είπα νωρίτερα ότι η Κομισιόν ε, πρότεινε την ε, υποχρεωτική ενδιάμεση αξιολόγηση και να υπάρχει τροποποίηση των τελευταίων ε, δύο ετών των προγραμμάτων. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι σαφές πώς θα αξιολογηθούν οι επιδόσεις καθώς τα κράτη-μέλη θα μπορούν να κάνουν σημαντικές μεταφορές πιστώσεων χωρίς έγκριση και έτσι θα αυξάνεται ο κίνδυνος ότι θα γίνουν τροποποίησεις χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα. Και αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα τη ένταση που συχνά υπάρχει μεταξύ τη επιθυμία των κρατών μελών να δαπανίσουν τα διαθέσιμα κονδύλια και τη ανάγκη να διασφαλίσουν ότι φυσικά οι δαπάνε οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα για του πολίτε. Αυτά για τη σημερινή μας δουλειά και εδώ κάποιες σύντομες πληροφορίες για τις ε, εκθέσεις ε, στο μέλλον, που θα πλησιάσουμε στο μέλλον από το τμήμα 2 τους επόμενους μήνες και έτη. Μπορείτε να δείτε ότι έχουμε τις ετήσιες εκθέσεις. Ε, θα έχουμε ε, ουσιαστικά μια, ένα νέο εγχείρημα για τις επιδόσεις, αλλά για τις εκθέσεις επιδόσεων θα δείτε ότι καλύπτουμε ε, την κινητικότητα, την αστική, την... τις ναυαρχίδες, στις μεταφορές, τις πολιτιστικές επενδύσεις, την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Αυτό είναι περίπου βιομηχανία 4.0, πολύ ενδιαφέρον ε, θέματα, διασυνορικά προγράμματα, την παιδική φτώχεια. Αυτό είναι τώρα για το έτος 2020 και για το επόμενο έτος έχουμε και πάλι διαφορά ενδιαφέροντα θέματα που μπορείτε να τα δείτε στη διαφάνεια. Ελπίζω να μπόρεσα να καλύψω όλα τα θέματα και εντό χρόνου. Και ανυπομονώ να ακούσω τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ιβάνοβα για την πολύ πλούσια παρουσίαση και στο προηγούμενο και στις συστάσεις. Θα ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση. Θέλω να χαιρετήσω και την παρουσία και του κύριου Βενμπρέσκα, που είναι διευθυντής της ΓΑΜΑ Δελταρίτζιο και θα μπορούσε να λάβει το λόγο στη συζήτηση για τα θέματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Να δώσω το λόγο στην Κωνστά Σκρέλ. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την παρουσίαση, η οποία ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Και για μένα η καλύτερη είδηση που ακούσαμε ήταν το ότι η πολιτική συνοχή παρουσιάζει επίπεδο ασφάλματο μόνο τη τάξη του 3%. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία γιατί αγωνιστήκαμε επί σειρά ετών ε, προκειμένου να μειώσουμε ακριβώ, να συγκνώσουμε αυτό το επίπεδο ασφάλματο. Και ελπίζω ότι η αναδιάρθρωση, αν θέλετε, του, ε, της ε, τάξης των οικονομικών με βάση ακριβώς τον κανονισμό Omnibus μας επέστρεψε να το επιτύχουμε μεταξύ άλλων. Μαζί δηλαδή και με τις προτάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη-μέλη και οι οποίες υλοποιήθηκαν από την πλευρά τους. με πλήση το γεγονός ότι υπάρχουν μία σειρά από αρμοδιότητες τις οποίες έχει αναλάβει το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν ήξερα, για παράδειγμα, ότι ελέγχεται και το τι ακριβώ κάνουμε σε επίπεδο ε, ε, εφαρμογή τη νομοθεσία και κατά πόσο τα όσα πράττουμε τελικά είναι χρήσιμα. Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι ε, εμεί ω Κοινοβούλιο και εγώ ω εισηγήτρια σε ό,τι αφορά το γενικό κανονισμό, δηλαδή των κοινών διατάξεων, εμ, καταφέραμε να συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο του στόχου μα Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, την καινοτομία, την καταπολέμηση τη ένδυα, Όλα λοιπόν αυτά τα ζητήματα, όλα αυτά τα θεματικά πεδία έχουν καταστεί πολύ σαφή και αναφέρονται τα μέσα στο κείμενο του νέου κανονισμού. Άρα λοιπόν αυτό που θα πρέπει τώρα να κάνουμε είναι να καταδείξουμε στα κράτη-μέλη πώς ακριβώς να εφαρμόσουν αυτά τα στοιχεία στην πράξη. Και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα. Τώρα σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση αναθεώρηση, το midterm review, νομίζω πως θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βρούμε τη χρυσή τομή, δηλαδή που να εξυπηρετήσει όλες τις πλευράς. Θεωρώ πως ε, από τη μία πλευρά χρειάζεται να υπάρχει απαραίτητη ευελιξία και σε αυτό έχετε δίκιο, ότι δηλαδή υπάρχει λόγος να διασφαλίσουμε αυτή την ευελιξία, αλλά από την άλλη πλευρά χρειάζεται να υπάρχει και κάποια ασφάλεια, μια σιγουριά σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, ειδικότερα σε ό,τι αφορά προγράμματα και project που τρέχουν επί σειρά ετών. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα δηλαδή στην ευελιξία και την σταθερότητα, την ασφάλεια του προγραμματισμού. Και εδώ με εξέπλησε λίγο το γεγονός ότι στο πεδίο που αναφερόταν ε, στην ε, τρέχουσα ε, περίοδο έχετε αναφέρει ως το αποθεματικό επιδόσεων βρίσκεται σε κίτρινο χρώμα, γιατί το αποθεματικό αυτό ήταν ουσιαστικά το χειρότερο το οποίο έχουμε κάνει στα τελευταία χρόνια στην πολιτική συνοχή, αφού ήταν απολύτως άχρηστο. Οπότε εδώ θα ήθελα το πεδίο δηλαδή να έχει κόκκινο χρώμα και όχι κίτρινο, αλλά εντάξει. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες ε, που κάνουμε, ε, καθώς αυτό που μας ενδιαφέρει όλους μας είναι να μπορέσουμε να οργανώσουμε στην πράξη μια καλύτερη πολιτική συνοχή για τις περιφέρειες και τις περιοχές. Ε, και αυτό που είπατε κι εσείς, δηλαδή ότι η απλούστευση των σχετικών ε, ε, των ε, σχετικών ισολογισμών και η, η, η, αξιολόγηση των κατά πόσο και με ποιον τρόπο δαπανώνται αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια παραμένουν βασικές προτεραιότητες. Αλλά ε, είναι σωστό και αυτό που είπατε και είναι πολύ χρήσιμο και μελλοντικά, δηλαδή να βρισκόμαστε σε τακτική επικοινωνία μεταξύ μας εδώ, με την Επιτροπή μας δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Βακόφ. Ο Ανδρέα Νούβακοφ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πάντα με χαρά μου ακούω τις παρουσιάσεις τη κυρίας Σεβανόβα εδώ ε, και η Κωνστάστα θα πρέπει να πω ότι ήταν ε, διπλωματική στην τοποθέτησή τη ο Συνήθω. και είναι θετικό βέβαια αυτό. Αλλά μετά από την παρουσίαση της κυρίας Βάνουα, θεωρώ πως εμεί ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ε, έναν ακόμα σύμμαχο στο πλευρό μα, ε, δηλαδή το Ελεκτρικό συνέδριο, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό κοινών τάξεων. Οπότε, εάν ε, θα μπορούσαμε να έχουμε την κυρία Ιβάνοβα μαζί μα στον επόμενο τριμερή διάλογο, θα μπορούσαμε να έχουμε καταλήξει σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει πριν από τα Χριστούγεννα. Είναι πολύ θετικό το γεγονό ότι κάνετε δουλειά τόσο σε βάθο, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το κομμάτι ακριβώ τη πολιτική συνοχή και ε, τα όσα κάνετε για την επόμενη προγραμματική περίοδο, ε, νομίζω πως ε, επιτελούνται ακριβώς στην κατάλληλη χρονική συγκυρία. Δηλαδή, μία από αυτές τις εκθέσεις μας είπατε ότι θα δημοσιευτεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Δηλαδή, ακριβώς την περίοδο εκείνο που θα αναλάβει η Κροατική Προεδρία και θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσει μαζί μας. Ε, το θέμα όμως είναι ότι χθες κάναμε μια συζήτηση ε, με το Γενικό Διευθυντή ε, Eurostat και ε, σήμερα κάνουμε μια συζήτηση μαζί σα σε ό,τι αφορά την πολιτική και πάλι συνοχή και τα στοιχεία και του αριθμού που έχουμε στη διάθεσή μα. Και γιατί το αναφέρω, γιατί υπάρχουν μια σειρά από άρθρα τα οποία κατακεραμνώνουν την πολιτική συνοχή και θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι δεν είναι υπέρ της πολιτικής συνοχής. Βασιζόμενος λοιπόν στα όσα μα λέτε και στα όσα έχουμε δει και επιτόπου, νομίζω πως μπορούμε να αποδείξουμε ότι πέραν από τους υπολογισμούς, θεωρητικό επίπεδο, τους μαθηματικούς υπολογισμούς και τους ισολογισμούς, δεν υπάρχουν κάποιοι, ε, εκείνοι δηλαδή οι οποίοι τελικά σε στελική ανάλυση συνεισφέρουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι αποφελούνται από την πολιτική συνοχή. Τελικά δηλαδή όλοι βγαίνουν κερδισμένοι από την ε, εφαρμογή της πολιτικής συνοχής ε, και νομίζω πως ε, μπορούμε από κοινού εδώ οι συνάδελφοι από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο να βρούμε ε, μια καλύτερη λύση για τη μελλοντική πολιτική συνοχή, χωρί όμω να την εξαλείψουμε. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τι προσπάθειε που κάνετε σε σχέση με την απλούστευση, θα πρέπει να πω πω είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Δηλαδή, θυμάμαι ε, στο δεύτερο έτο τη πρώτη μου θητεία εδώ στο Κοινοβούλιο είχαμε ξεκινήσει την συζήτηση του κανονισμού για την απλούστευση και είχαμε ξεκινήσει το σχετικό διάλογο και υπήρξε και μια έκθεση 50 σελίδων η οποία μας ανέφερε το πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτή την υπεραιτέρω απλούστευση. Ε, δεν μπορώ όμως να, να θεωρήσω ότι οι δικαιούχοι ε, στα δεύτερα κατημέλια αντιλαμβάνονται τι, τι ακριβώς θέλουμε να επιτύχουμε από όλα αυτά. Πάντως, ε, ε πρόσφατα συζητήσαμε εντατικά και με πάθο ε, το e-cohesion, δηλαδή την ε, συνοχή, του πώς αυτή την πολιτική συνοχή πώς εφαρμόζεται σε ηλεκτρονικό επίπεδο. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε, εσείς δραστηριοποιείστε ως ελεκτικό συνέδριο και σε αυτό το τομέα του e-cohesion και πώς ε, θα μπορούσε δηλαδή να επηρεάσει την απλούστευση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των κοντιλίων τη πολιτική συνοχή. Γιατί θα πρέπει να πω ότι το ποσοστό απορρόφηση των κοντιλίων τη σήμερα ημέρα είναι απογοητευτικό. Δηλαδή μόνο 33%. Οπότε ακριβώς το eco θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τους τρόπους μέσω των οποίων μέσα στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα επιτύχουμε υψηλότερη απορρόφηση των κοντιλίων. Thank you ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Ιβάνοβα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Αλλά θα θέσω το ερώτημά μου στα φιλανδικά, αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε. Ναι, Κύριε Αβάνοβα, η έκθεσή σας είναι πολύ ενδιαφέρουσα και εγώ τη διάβασα. Και διαπίστωσα ότι περιλαμβάνει μία σειρά από χρήσιμε πληροφορίε ε, για του σκοπού μα, ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή το μέλλον τη πολιτική συνοχή. Αλλά θα ήθελα να εκφράσω και μία ευχή το μέλλον. Κατά τη δική μου άποψη λοιπόν και με βάση τη δική μου εμπειρία θεωρώ πως ε, είναι πολύ σημαντικό ε, σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής να λαμβάνουμε όσο το δυνατόν ποιοτικότερα δεδομένα σε ό,τι αφορά ακριβώς αυτό τον αντίκτυπο ε, που είχε πολιτική συνοχή και στο παρελθόν γιατί υπάρχουν κάτι μέλη τα οποία λαμβάνουν από τα κονδύλια της, ε, από τα δηλαδή μέτρα της πολιτικής συνοχής 20 ευρώ ανά πολίτη. Αλλά σε άλλα κράτη-μέλη αυτό το ποσό ανέχεται σε 360 ευρώ κατά κεφάλι δηλαδή ετησίως. Οπότε είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο είναι ο αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής στα επιμέρους κράτη-μέλη, στις διαφορετικές περιοχές και περιοχέ με βάση δηλαδή την ταξινόμηση ΝΑΤΣ. Ειδικότερα αναφέρομαι στι ΝΑΤΣ 2 και ΝΑΤΣ 3. Και αναφέρομαι δηλαδή στις διαφορές που υπάρχουν ακριβώς στην ένταση των ενισχύσεων, γιατί υπάρχει χαμηλή ένταση ενισχύσεις σε ορισμένες περιοχές, υψηλότερη σε άλλες. Οπότε ε, θεωρώ πως θα έχετε ε, δεδομένα σε συγκεκριμένες χρονικές σειρές, τα οποία θα μπορούσαν να μας φανούν χρήσιμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Μουτζανόφσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω, όπως οι προθυλαλήσατε στην ομολήτρια, για την ακρίβεια των δεδομένων που μας παρουσίασε και είναι μια πολύ σημαντική περίοδος αυτή για την ε, πολιτική συνοχής. Η δουλειά μας στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι πράγματι πολύ ουσιώδες και πολύ σωστά το έθεσε ο πρόεδρος της Επιτροπής μας. Με μεγάλο ενδιαφέρον ε, σας άκουσα να μιλάτε για την απλούστευση των ελέγχων, για την αρχή της ευελιξίας επίσης πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για να δαπανίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κονδύλια στο πλαίσιο των ε, δημοσιονομικών προοπτικών και του παρελθόντος και του παρόντος και του μέλλοντος. Σαφέστατα τα επίπεδα σφαλμάτων, το error rate, είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και πρέπει να δούμε και πώς ε, δαπανούν τα κράτη-μέλη ε, τα χρήματα σε σχέση με τους στόχους για να βελτιώσουν την καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη ακρίβεια των δεδομένων, η ανάλυση, η λεπτομέρεια είναι αυτά που βάζουν τις βάσεις για σωστή συνεργασία έτσι ώστε να σχεδιάσουμε και να αξιοποιήσουμε την πολιτική συνοχής και να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Αυτό θα ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ολμπράιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω τρία ερωτήματα να σας θέσω. Ένα για το παρελθόν και δύο για το μέλλον. Ως προς το παρελθόν. Στην Επιτροπή Κοντ ε, θα ασχοληθούμε με τα επίπεδα σφάλματος. Είναι πολύ σαφής αυτή η πληροφόρηση για εμάς. Γιατί το επίπεδο σφάλματος είναι ψηλότερο από πέρσι, φέτος. Και αν αυτό το συνδυάσουμε με ε, τη ε, στοιχεία του Διευθυντή Λεμέτχο, ο οποίος λέει ότι ο ρυθμός υλοποίησης είναι πολύ χαμηλός, κάτι που έχει υποθεί σε αυτή την Επιτροπή. Όταν λοιπόν συνδυάζουμε τη χαμηλή υλοποίηση συν το υψηλό επίπεδο σφάλματος, τίθεται το εύλογο ερώτημα, μα τι συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη συζήτηση που θα έχουμε για την πολιτική συνοχή. Επίσης, στην παρουσίασή σας παρουσιάσατε από κοινού το παρελθόν με το μέλλον. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή για ελεγκτικό συνέδριο. Όμως, ως προς το μέλλον, κάτι που μας ενδιαφέρει είναι το εξή. Τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε έχουν να κάνουν με δυνάμει περικοπές σε θέματα κονδυλίων συνοχής για κάποια κράτη-μέλη και δεν είναι αυτά τα νούμερα που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο του 2018. Μείον 23% παρουσιάστηκε για την Πολωνία το Μάιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ στη δική σας έκθεση ήταν μείον 19% για την Πολωνία. Μπορεί να έχω σφάλει βέβαια. Αλλά εν πάση το ερώτημα άμα αφορά τα αριθμητικά στοιχεία, τα νούμερα, τι άλλαξε μεταξύ 18 και 19 για να έχουμε υψηλότερο επίπεδο σφάλματος. Θέλουμε να καταλάβουμε την νοοτροπία. Δεν το θέμα οι περικοπές, αλλά η αλλαγή της πολιτικής συνοχής και αυτό είναι σαφέστατο. Και τελευταίο ερώτημα ως ελεγκτικό συνέδριο. Πώς συγκρίνεται τα στοιχεία για την πολιτική συνοχή με, την, ε, με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες αφού δεν υπάρχουν προτεραιότητες ή θα πάρετε τη θεματική συγκέντρωση ως προτεραιότητα. Δηλαδή, δεν έχουμε ευρωπαϊκή στρατηγική, αλλά έχουμε θεματική συγκέντρωση αναθεματικούς άξονες, να το πω έτσι. Αυτό το θεωρείται ευρωπαϊκή προτεραιότητα ή όχι. Ή λέτε αυτό που είπατε ότι εμείς ως ελεκτικό συνέδριο σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία ε, στρατηγική. Έχει σημασία για μένα που είμαι εισηγητής για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η στρατηγική θα είναι αποτέλεσμα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαίσιου. Άρα το πι θα είναι η στρατηγική. Θα έχουμε στρατηγική έπαξη και δούμε τα νούμερα. Πώς θα θέλατε δηλαδή να τοποθετηθείτε στο μέλλον και προς τα που θα κινηθείτε. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. La question de... Ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημα του κυρίου Γιάνν Ολμπράιντ είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί μπορεί να αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ συναδέλφων. Και θα ήταν και για μας ενδιαφέρον να ακούσουμε το ελεκτικό συνέδριο να επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει στρατηγικό όραμα. Το συζητήσαμε χθες. Και έχεις Απόλυτο δίκιο και πολύ καλά κάνεις που θέτεις αυτό το ερώτημα. Οι θεματικοί στόχοι αποτελούν στρατηγικό όραμα ή όχι. Είναι πολύ πολιτικά αυτά τα ερωτήματα και θα πρέπει να τα συζητήσουμε εμείς μεταξύ μας επίσης, διότι αυτό παραπέμπει στο δικό μας πλαίσιο του CPR, το κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Είναι ένα έγγραφο αυτό το οποίο εντάσσεται σε συγκεκριμένο πολιτικό όραμα. Είναι θεμελιώδες το ερώτημα. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ιβάνοβα να απαντήσει. Θέλω επίσης να πω ότι ενδεχομένως να μην υπάρχει άλλη πολιτική που να έχει μετρηθεί τόσο όσο η περιφερειακή πολιτική. 9.000 δείκτες μου έχετε πει ότι υπάρχουν ή έχουν υπάρξει που επιτρέπουν την αξιολόγηση των επιδόσεων αυτής της πολιτικής. Είναι μια πολιτική λοιπόν η περιφερειακή πολιτική που ελέγχεται εξαιρετικά πολύ και μπορούμε πράγματι να πούμε ε, ε, κατά πόσο αποδίδει αν έχει επιδόσεις ή δεν έχει. Και υπάρχουν και πάρα πολλές επικρίσεις για την πολιτική συνοχής, τις οποίες υπογραμμίσατε κι εσείς, που δείχνουν ε, τις ανεπάρκειες άλλων πολιτικών, γιατί η πολιτική συνοχή ε, εφαρμόζεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο απουσιάζει, από το οποίο απουσιάζει η συνοχή και με συστηματικό τρόπο υπενθυμίζουμε την ανάγκη να υπάρχει συνοχή μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών πολιτικών. Επομένως, πριν σας δώσω το λόγο, θέλω και εγώ να σας θέσω ένα δικό μου ερώτημα, που έχει να κάνει με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Εισαγγελικής Αρχής. Κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να συνεργαστεί η Eurojust με την Olaf, με τη Frontex και τη Europol και την Εισαγγελική Αρχή, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ποιος είναι ο ρόλος του ελεγκτικού συνεδρίου σε αυτή τη συστάδα, σε αυτό το συσχετισμό και πώς ε, περιμένετε να εξελιχθεί η συνεργασία σας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και σας θέτω αυτό το ερώτημα, διότι Έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο όπου υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις ενίοτε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής εισαγγελία στην πολιτική συνοχή. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δέχθηκε ξεκάθαρα πάρα πολλές επικρίσεις με τις παρεμβάσεις των ΜΕΝ και των ΔΕ Άρα, αν συμφωνείτε, να δώσουμε συντομία το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στις επικρίσεις που δέχθηκε και μετά θα έχετε εσείς το λόγο για να μας δώσετε τις απαντήσεις σας. Κύριε Διευθυντή, ε, σας ακούμε. And also Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ την προσεκλημένη μας και την ομάδα μας για όλες αυτές τις εκθέσεις. Θα είμαι πολύ σύντομα σε ένα από τα ερωτήματα που ανακύψαν γιατί υπάρχει υψηλότερο επίπεδο σφάλματος θα πρέπει να δώσω το λόγο στο συνάδελφο, στη συνάδελφο από το τμήμα ελέγχων της ΓΔ Ρίζιο, γιατί γνωρίζει καλύτερα. Εγώ θα είμαι σύντομος. Ε, προέκυψε το θέμα της εκδομική ε, συνοχή είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της πρότασής μας. Πιστεύουμε ότι όλη η ανταλλαγή δεδομένων στο μέλλον θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά αυτό θα οδηγούσε σε τρομερή μείωση του διοικητικού άχθους για τους δικαιούχους. Επίσης, θα είμαστε πρόθυμοι να βρούμε μια συμφωνία με τους συνομοθέτες, γιατί κατανοούμε εδώ ότι το πρόβλημα περισσότερο έγινε στο Συμβούλιο και όχι στο Κοινοβούλιο και πρέπει να βρούμε τρόπους ε, για το πώς οι διαχειριστές των προγραμμάτων μπορούν να βοηθήσουν τους δικαιούχους όχι μόνο προωθώντας την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων αλλά και βοηθώντας τους ε, στην ψηφιοποίηση αν χρειάζεται. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό για μας, ε, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε σημαντικά κέρδη εδώ και μείωση του διοικητικού άχθους. Το δεύτερο θέμα, συμφωνούμε πολύ σημαντικά με την κυρία Κρέλ εδώ, ότι η σημερινή εκδοχή του ε, αποθυματικού επιδόσεων ε, είναι ιδιαίτερα μηχανική, δεν είναι φυής. Θα πρέπει να μεταφέρουμε χρήματα αν δεν πετυχαίνουμε κάποιους στόχους. Αυτό έχει υποθεί εδώ και χρόνια και μερικές ε, φορές δεν είναι στον έλεγχο των διαχειριστών των προγραμμάτων. Γι' αυτό πιστέψαμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε ε, το σημερινό αποθεματικό επιδόσεων και να το διατηρήσουμε έτσι, γιατί θα έχουμε μια ενδιάμεση αναθεώρηση. Αλλά επίση να εισαγάγουμε και κάποια ευελιξία, γιατί στην ε, σημερινή προγραμματική περίοδο είδαμε ότι όταν είχαμε την μεταναστευτική κρίση είχαν προγραμματιστεί όλα τα χρήματα και δεν, υπήρξε, δεν υπήρχε δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει με κονδύλια τη πολιτική συνοχή και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε στον εαυτό μας κάποια ευελιξία και ενώ, όπως είπε η κυρία Κρέλ, θα σεβόμαστε και την απαραίτητη σταθερότητα για τα μακροπρόθεσμα προγράμματα, αλλά τουλάχιστον να έχουμε κάποια ευελιξία για την αντιμετώπιση και νέων προκλήσεων. Και τέλος, θα αναφερθώ στην απλούστευση. Πιστεύουμε το μεμονωμένο μεγαλύτερο πρόβλημα της πολιτικής συνοχής είναι η πολυπλοκότητά της σήμερα. Και γι' αυτό προτείναμε 80 ε, μέτρα πλούστευσης ε, και περισσότερο ενισχύω ότι πολλά από αυτά τα μέτρα θα αποδυναμωθούν στη συζήτηση. Και αυτό που θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε είναι να είναι δυνατόν πιο απλά τα πράγματα για τους δικαιούχους. Και αν μπορώ να δώσω το λόγο στον συνάδελφο για να πει μια-δυο προτάσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι πολύ σύντομο. Συγγνώμη, είδωσα το λόγο στην Κομισιόν για μία παρέμβαση. Αλλά να δώσουμε το λόγο στην εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους αξιότιμους βουλευτές. Νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω και στην ερώτηση της Κομισιόν, γιατί η απάντηση είναι περίπου ίδια και είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Ευχαριστώ τον κύριο Όλμπριχτ. Μάλιστα ήταν η πρώτη ερώτηση που το 3% αλλά ήταν το προηγούμενο έτος. Φέτος έχουμε 5%. Και η ερώτηση είναι γιατί έχουμε ανώτερο επίπεδο από το 3% που ήταν το περασμένο έτο. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Καταρχήν, να πω το εξή. Θα το έθετα ω εξή. Δεν είναι ότι φέτος έχουμε ένα συνήθιστο επίπεδο σφάλματος, αλλά μάλλον πέρσι είχαμε συνήθιστα χαμηλό επίπεδο σφάλματος. Ο κύριο λόγος ήταν ότι είχαμε πολύ χαμηλό ποσοστό πληρωμών. Είχαμε μόνο 80 δισεκατομμύρια πληρωμών στι δαπάνε, ενώ αν το συγκρίνουμε με φέτος έχουμε πάνω από 23 δισεκατομμύρια πληρωμών. Συνήθω όταν έχετε χαμηλότερες, χαμηλότερο ποσοστό πληρωμών, τότε θα είναι χαμηλότερο και το επίπεδο σφάλματο. Επίσης, στο δείγμα του τελευταίου έτους είχαμε ε, πολύ μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών μέσων στο δείγμα, ενώ φέτος ε, είχαμε περισσότερα είδη λαθών, ε, κάποια προγράμματα που δεν ήταν επιλέξιμα, δαπάνες που δεν ήταν επιλέξιμες, προβλήματα στις δημόσιες συμβάσεις. Βέβαια, δεδομένου του υψηλότερου ποσοστό, ε, του, μεγαλύτερου ποσού, άνω του 23 δισεκατομμύρια, είναι υψηλότερο και το επίπεδο ασφαλίματο. Και θα σύγκρινα αυτό το 5% με το προ-προηγούμενο έτους, όπου είχαμε 4,8%. Έτσι λοιπόν αυτό μπορεί περισσότερο να συγκριθεί με το 4,8 και πιο σταθερό αν θέλετε. Σίγουρα δεν είναι κάτι θετικό, αλλά είναι πιο σταθερό σε σύγκριση με το περσινό 3% που ήταν ε, εξαιρετικά χαμηλό. Και του χρόνου θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί θα είναι υψηλότερο το επίπεδο σφάλματος. Αλλά όπως σας είπα, επειδή είχαμε χαμηλότερο επίπεδο δαπανών. Χαμηλότερο, ε, χαμηλότερο ποσό δαπανών. Λοιπόν, Ξεκινάω με την ερώτηση του κυρίου Όλμπρικτ για τις ε, διαφορές ε, στα ποσοστά. Δεν θα ανησυχούσα και τόσο γιατί ο σκοπός εδώ δεν είναι αυτός. Παρουσιάσαμε τις πληροφορίες τη στιγμή που τις είχαμε, τη στιγμή που δημοσιεύτηκε το έγγραφο. Φυσικά αλλάζουν τα πράγματα. Είχαμε μεταβολή. Στη συνέχεια όμως εδώ η κύρια ιδέα της επισκόπησης είναι να δείξουμε τη φιλοσοφία, το πώς γίνεται η προκατανομή, πόσο διαφανής είναι η διαδικασία. Φυσικά δεν είχαμε τα εργαλεία και το χρόνο να ελέγξουμε τι συμβαίνει στα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Ο στόχος είναι πιο φιλοσοφικός, να εξηγήσουμε τι σημαίνει η διαδικασία της προκατανομής, ποια είναι τα νέα στοιχεία και να δείξουμε ότι έχουν υπάρξει βελτιώσεις στη διαφάνεια, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν πολύπλοκα τα πράγματα. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα νομίζω εδώ παρά οι διαφορές ε, στα νούμερα. Αλλά για την άλλη σας ερώτηση για τη στρατηγική. Πραγματική, για μένα είναι η πιο σημαντική ερώτηση και σας ευχαριστώ που μου θέτετε την πρόκληση αυτή. Δεν μπορώ να πω παραπάνω από όσα είπα και δεν θέλω τώρα να λάβω πολιτική θέση γιατί το ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι πολιτικό όργανο. Απλώς ε, αναφέρουμε τα γεγονότα, κάνουμε κάποιες συστάσεις ε, και εξάγουμε συμπεράσματα, όμως οι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται από εσά. Και ελπίζω ότι ε, θα μπορούσα να σας βοηθήσω τα γράφα αυτά να λάβετε τις κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις, αλλά δεν υπάρχει στρατηγική σε σύγκριση με το είδος ε, της στρατηγικής που είχαμε στο Ευρώπη 2020. Αυτό λέμε. Δεν υπάρχουν θεματικές συγκεντρώσεις φυσικά στο CPR. Υπάρχει ένας κατάλογος στόχων και υπάρχουν και διάφοροι άλλοι στόχοι που αναφέρονται εδώ και εκεί, όπως σας είπα, διάσπαρτα. Όμως, ε, όταν ε, προσπάθησα εγώ να εξετάσω και ζήτησα και την Κομισιόν ε, Πολάκης να μας παρουσιάσει ένα συνεκτικό έγγραφο που να μπορεί να συγκριθεί με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, με κατεύθυναν στις διακηρύξεις Μπρατισλάβα και Ρώμης. Αυτά τα δύο έγγραφα δεν συγκρίνονται, δεν είναι συγκρίσιμα. Με συγχωρείτε αλλά το ένα είναι ένα φύλλο χαρτί και το άλλο είναι δύο-τρεις σελίδες, αλλά δεν μπορούν να συγκριθούν με τους μετρήσιμους συγκεκριμένους στόχους που θα θέλαμε να πετύχουμε, πριν το σχάρι ε, τις ομάδες στόχους, συγκεκριμένους στόχους. Αν δεν τους έχεις αυτούς, τότε αργότερα θα είναι πολύ πιο δύσκολο να είναι αν έχει πετύχει κάτι, αν δεν μπορεί να το μετρήσει σε σχέση με έναν αρχικό στόχο, σε σχέση με μια αρχική στρατηγική που μπορεί να είχε. Αυτή είναι η απάντησή μου και συγγνώμη που δεν μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένη. Σα ευχαριστώ για την ερώτηση πάντω. Και να έλθω τώρα στι ερωτήσει τη κυρία Κρέλ για το επίπεδο σφάλματο. Νομίζω απάντησα γιατί δεν έχουμε 3 αλλά 5% και για την υψηλότερο. Για την περίπτωση τη προτάσει Κομισιόν. Ναι. Αυτά τα έγγραφα τα δημοσιεύουμε ως γνωμοδοτήσεις. Ελπίζουμε ότι θα είναι χρήσιμα σε εσά για να λάβετε τις αποφάσεις, κυρίως όταν παρουσιάζονται εγκαίρως, για να σας βοηθήσουν στη διαδικασία διαπραγματεύσεων. Ελπίζω λοιπόν ότι η γνωμοδότηση για το CPR θα είναι χρήσιμη, αν και είναι κάπως παλιά, όπως σας είπα. Για την ενδιάμεση αναθεώρηση και το να βρούμε κοινοτόπο, συμφωνώ και για την ευελιξία και για το σχέδιο να πετύχουμε την ισορροπία και μάλιστα την ε, ισορροπία μεταξύ απλούστευσης και ελέγχου. Αυτό είναι ένα θέμα που πάντοτε το τονίζαμε. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Τώρα, ε, γιατί δεν ήταν κόκκινε οι επιδόσει. Ε, εξακολουθούμε να έχουμε πολλά κόκκινα, ρωτήστε την Κομισιόν. Δύο έχουμε, αλλά και πάλι είναι πάρα πολλά. Αλλά αφού αξιολογήσαμε και τι 14 κατευθυντήριε αρχέ είδαμε ότι η Κομισιόν κάλυψε όλα τα βήματα που είχαν ληφθεί και θεωρούμε ότι σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να δώσουμε κίτρινο χρώμα. Βέβαια υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης, περιθώριο βελτίωσης πάντοτε υπάρχει. Και σας ευχαριστώ κύριε Νόβακοφ που είπατε ότι είναι χρήσιμο το έργο μας. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμη και αν βρήκατε κάποια θετικά μήνυματα, εμεί ω Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο ε, δεν υπερασπίζουμε τι πολιτικέ συνοχέ. Ε, μην ε, μα παρανοήσετε. Εδώ απλώ θέλουμε να παρουσιάσουμε την αντικειμενική εικόνα και την αντικειμενική άποψη βάσει των γεγονότων. Όπου βλέπουμε ελλείψεις, τις τονίζουμε. Όπου βλέπουμε θετικές εξελίξεις, προσπαθούμε να τις παρουσιάσουμε λίγο και περισσότερο. Ίσως αυτό είναι το καινούριο, που προσπαθήσαμε να δείξουμε περισσότερο τις βελτιώσεις, αλλά ας μην ξεχνάμε και τα προβλήματα που έχουμε. Το επίπεδο σε τη εξολοκουθεί να είναι πάνω από το 2%, εξακολουθεί να είναι υψηλό. Παρ' όλα αυτά. Είχαμε σημαντικές βελτιώσεις ε, από τα έτη 2000-2007 όταν είχαμε ε, επίπεδο σφάλματος 11-12%. Ε, Τώρα έχει πέσει, αλλά και πάλι είναι πάνω από το 2%. Το 2% είναι το ελάχιστο κατόφλι. Αυτό θεωρούμε το ελάχιστο επίπεδο. Έτσι λοιπόν εξακολουθεί να πρέπει να γίνει κάποια δουλειά εκεί για το αντίκτυπο και τα αποτέλεσματα της συνοχής και τα καλά δεδομένα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική ερώτηση που τέθηκε για την ποιότητα των δεδομένων. Και εδώ βασιζόμαστε στην Κομισιόν, κυρίως ε, σε ό,τι αφορά τη ε, νέα διαδικασία πιστοποίησης. Αν δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τα δεδομένα και να βασιστούμε στα δεδομένα και στη δουλειά άλλων, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτή τη νέα προσέγγιση. Αυτό είναι σημαντικότατο στοιχείο να έχουμε καλά στοιχεία, καλά δεδομένα. Ε, φυσικά δεν έχετε καλούς δείκτες, δεν μπορείτε και να μετρήσετε. Σε αυτό επενερχόμασταν στις 14 ε, κατευθυντήριες αρχές. Για την απλούστευση, νομίζω ήδη απάντησα. Τα ακριβή δεδομένα επίσης αναφέρθηκαν από την κυρία Μεζανόφισκα. Σύμφωνα απόλυτα μαζί σας. Θα πρέπει να μπορούμε να μετράμε με τους σωστούς δείκτες και να απλουστεύουμε. Όχι μόνο χάρη της απλούστευσης, αλλά να έχουμε και ένα σκοπό, να υπάρχει ένα νόημα και να διατηρούμε πάντοτε την ισορροπία. Για τη δική σας ερώτηση, Πρόεδρε, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν μπορώ να πω πολλά φοβάμαι. Πριν να έχει διοριστεί το πλήρες σώμα στην εισαγγελία, και να αναλάβει καθήκοντα, αλλά μπορώ να σας πω ότι σε όλα τα επίπεδα είχαμε ήδη μια σχετική παρουσίαση από τις υπηρεσίες του στο Λουξεμβούργο για το πώς αναμένουν να οργανωθεί η δουλειά τους και εμείς από τη δική μας πλευρά είμαστε ανοιχτοί και επιδεικνύουμε πνεύμα συνεργασίας. Εμείς ως ελεκτικό συνέδριο δεν προβαίνουμε σε ερευνές ε, για περιπτώσεις απάτης. Υπάρχει πολύ σαφή διάκριση ε, καθηκόντων. Ε, φέτος είχαμε 9 υποθέσεις που παραμέψαμε στην Όλαφ. Αυτή είναι η υπηρεσία που προβαίνει στις ε, έρευνες. Αλλά όταν εντοπίζουμε τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιες υποθέσεις, δεν ξεκινάμε εμείς οι ίδιοι τις διαδικασίες, αλλά τις παραπέμπουμε τις υποθέσεις αυτές στην Όλαφ και έχουμε πολύ καλή συνεργασία μαζί τους. Φαντάζομαι ότι αυτό θα ισχύει και με την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις που δώσατε. Ήταν πολύ πλούσια η σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ και πάλι τους συναδέλφους ε, για την ποιότητα των ε, σχολείων τους και θέλω να σας πω στο επανειδή καλώς, καθώς ε, θα ξαναβρεθούμε σύντομα για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Και πάλι ευχαριστώ. Τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ενός λεπτού για να μπορέσει να αλλάξει εδώ το πάνελ γιατί σε λίγο θα έχουμε μια πολύ σημαντική στιγμή. Θα υποδεχτούμε τον πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών. Συνεχίζουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Έχουμε την ε, χαρά να ευχαριστούμε σήμερα τον κύριο Καλ Χάινς Λάμπερτ, τον πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, ε, που συνεργάζεται με τη δική μας Επιτροπή. Έχουμε πολύ στενές σχέσεις ε, εδώ και πάρα πολύ καιρό και φυσικά καλούμαστε σε κάτι τέτοιο λόγω της ε, καλής λειτουργίας των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αγαπητέ Κάρλ, στο Παλέρμο ε, μας είπες ότι θα βλεπόμαστε. Η αλήθεια είναι, θα απόδειξη αποτελεί η σημερινή συνάντηση και θέλω να πω πόσο πολύ εκτίμησα το ρόλο που έπαιξε η Επιτροπή των ε, Περιφερειών, πόσο καλά μας υποδεκτήκατε και εμένα τον ίδιο προσωπικά στην εβδομάδα των Επιτροπών, των ε, Περιφερειών, με συγχωρείτε, και θα ήθελα να σου πω ότι εκτιμούμε πάρα πολύ τη δουλειά που έκανες ε, τα δύο τελευταία έτη από τότε που ανέλαβες επικεφαλής της Επιτροπής των Περιφερειών. Υπερασπίζεις ένθερμα τη συνοχή και το, του προγράμματος που έχετε ξεκινήσει πριν να ξεκινήσουν ε, οι διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, τυχαίνουν υποστήριξη από όλε τις περιφέρειες της Ευρώπης. Και θέλω να σου πω πόσο χρήσιμο μας ε, είναι αυτό στον κοινό αγώνα που δίνουμε σήμερα για να υπερασπίσουμε τη συνοχή και έναν πραγματικό προϋπολογισμό για τη συνοχή. Κατά την εβδομάδα των περιφερειών ε, εμείς συνεχίζαμε να απευθύνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη να μην θυσιάσουν τις παραδοσιακές τους πολιτικές και να μην θυσιάσουν την περιφερειακή πολιτική, την οποία χρειαζόμαστε πάρα πολύ σε όλη την Ευρώπη. Όμως, εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειαζόμαστε πάρα πολύ την Επιτροπή των Περιφερειών και χρειαζόμαστε να έχει έναν ενεργό ρόλο τα μέλη της να μπορούν ε, να ε, πιέζουν ε, τα κράτη-μέλη όταν λαμβάνουν χώρα ή διαπραγματεύσεις για το μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κυρία Καρλ Χάινς Λάμπερς, θα σας δώσω το λόγο για 15-20 λεπτά για να μας παρουσιάσετε τις σκέψεις σας για την πολιτική συνοχής, το πώς θα την υπερασπίσουμε αλλά να μας παρουσιάσετε και τα σημεία κλειδιά που θα πρέπει να υπερασπιστούμε στις ε, τρέχουσες διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα διάφορα ταμεία. Και θέλω να απευθυνθώ στους εισηγητές και στους ε, συνσηγητές ε, για τα διάφορα ταμεία. Εμείς γνωρίζουμε την ποιότητα της δουλειάς που έχει γίνει από τον εισηγητή της Επιτροπής ε, των Περιφερειών επί το συνόλου των κανονισμών και θέλουμε να επωφεληθούμε και να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και φυσικά έχουν ανοίξει ε, και ε, νέα θέματα, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ε, μετάβαση των ε, περιοχών ε, με λιγνίτη προς το να πετύχουν την ενεργειακή μετάβαση αυτή. Και αυτά αποτελούν έμπνευση φυσικά και για τη δική μας Επιτροπή για να προχωρήσουμε και στις δική μας εργασίες ως συνομοθέτες. Με μεγάλη χαρά σας δίνω το λόγο για 15-20 λεπτά και όλοι είναι υπομονούμενοι να σας ακούσουμε. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να παρουσιαστώ ενώπιόν σας σήμερα και να συμμετάσχω στις ε, εργασίες σας. Η συμμετοχή στις εργασίες σας καταδεικνύει όχι μόνο την εξαίρετη συνεργασία που σωστά υπενθυμίσατε είχαμε στο παρελθόν μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών, των αρμοδίων επιτροπών των δύο θεσμικών μας οργάνων, αλλά δείχνει η συμμετοχή μου στις εργασίες σας και ε, το μέλλον και τις προοπτικές για μια ιδιαίτερη έντονη και επικοδομητική συνεργασία μεταξύ αμφότερων θεσμικών οργάνων. Η πρώτη σας μετακίνηση εκτός έδρας είχε να κάνει με τη συμμετοχή σε μια εκδήλωση της Συμμαχίας για τη Συνοχή που έλαβε χώρα εντός της Επιτροπής των Περιφερειών ήταν μια ισχυρή πολιτική χειρονομία αυτή που εκτίμησαν ιδιαίτερω τα μέλη μας και το σύνολο των περιφερειών και πόλεων που συνεργάζονται και έχουν σφυριλατήσει τη συγκεκριμένη συμμαχία. Σήμερα το να εργαζόμαστε μαζί, να συνεργαζόμαστε είναι περισσότερο αναγκαίο παραποτέ γιατί περασπιζόμαστε κοινού στόχου ε, μπροστά και απέναντι σε εκπροσώπους κρατών μελών που επιδεικνύουν ευρωπαϊκή φιλοδοξία κάπως ισχυμική θα έλεγα και μπροστά στις προκλήσεις που οφείλει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη σήμερα. Και αυτό είναι και το νόημα του καθήκοντός μας. Το καθήκον μας είναι να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες του Ευρωπαίου πολίτη και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του. Οι προκλήσεις είναι πολυάριθμες και πολύ γνωστές θα έλεγα. Αυξάνονται οι ανισότητες, υπάρχει κλιματική αλλαγή. Φτωχαίνει η βιοσφαίρα και η βιοπικιλότητα. Έχουμε ε, διαχείριση μεταναστευτικής κρίσης και διαχείριση κρίσης ασφάλειας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φοντερ Λάιεν, πρότεινε τις έξι πολιτικές προτεραιότητες τις οποίες έχουμε μάθει πια σχεδόν απ' έξω όλοι. Και νομίζω ότι είναι σωστές οι προτεραιότητες αυτές. Όμως, θα πρέπει να δούμε πώς θα τις εφαρμόσουμε. Ενδιαφέρουσα μπορεί να είναι η ορολογία, αλλά μικρό επιχειρησιακό ενδιαφέρον. Η ευρεία συνένεση που επικρατεί σε σχέση με αυτούς τους στόχους θα πρέπει να αποτελέσει και το ισχυρό σημείο στην εκκίνησή μας. Είναι πολύ γνωστοί λοιπόν οι στόχοι και τους μοιράζονται όλοι. Ωστόσο, όταν γίνεται λόγος για τα μέσα επίτευξης των στόχων, εκεί αποκλίνουν οι απόψεις. Άλλωστε υπάρχει και το γνωστό ρητό που λέει ότι όταν, γίνεται, όταν μπαίνει το χρήμα στη μέση η φιλία διαλύεται. Η ψήφος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ισχυρή πλειοψηφία στις 10 του περασμένου Οκτωβρίου ενός ψηφίσματος που επιβεβαιώνει τους φιλόδοξους στόχους για το πολιετές δημοσιονομικό στέχιο καταδεικνύει του λόγου το αληθές όλων αυτών των πραγμάτων. Έχουμε το στόχο του 3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της Ένωσης των 27 και αυτό επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά από τις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις το βρίσκω πολύ σημαντικό. Αυτό που δημιουργεί πρόβλημα σήμερα είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Ο καθένας ή πολλοί έχουν ε, ε, ε, αιμονή με την έννοια της δίκαιης επιστροφής σε βάρος του ευρωπαϊκού συμφέροντος και της δίκαιης απόδοσης σας, της συνεισφοράς τους αν θέλετε. Και αυτό είναι πολύ θλιβερό ως συζήτηση. Ο Επίτροπος Έτιγκερ έχει εξηγήσει τη σημασία της τιμής του καφέ Δηλαδή έχουμε πει επανειλημμένο στο δημόσιο λόγο ότι αυτά που πληρώνει ο Ευρωπαίο πολίτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούν με ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα. Όμω, είναι καλύτερο να μιλούμε για τους καθαρούς αποδέκτες. Το να μιλούμε για τους καθαρούς αποδέκτες και τους καθαρούς εισφέροντες είναι κάτι το εντελώς απαξιωμένο πια και δεν είναι προς όφελος κανενός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προς όφελος όλων των χωρών. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα πρέπει να προασπιστούμε τα εθνικά συμφέροντα, όμως αυτά τα εθνικά συμφέροντα δεν μπορούμε να τα πειρασπιζόμαστε ε, ε, ως αντιτιθέμενα στα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Γιατί δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε ποιοι είναι πια οι καθαροί εισφέροντες και ποιοι είναι οι καθαροί αποδέκτες. Δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε για κάθε ένα από τα κράτη-μέλη τα ωφέλη π.χ. του Ευρωπαϊκού Διοδορυφόρου, ε, των ε, διασυνοριακών μεταφορών, τα ωφέλη των εξωτερικών συνόρων των κοινών. Και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε πόσο ωφέλει σε κάθε μία από τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ τυχή η ψή χώρα ξεχωριστά. Εξού και λέω ότι τα συμφέροντά μα είναι κοινά. Πρόσφατα είδα το μετρό τη Σόφια, ένα τεράστιο έργο που εκτελήσεται αυτή τη στιγμή, το οποίο στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας ε, έδωσαν ένα κατάλογο των δικαιούχων. Των δικαιούχων. Ποιες ήταν οι επιχειρήσεις, γερμανικές και άλλες. Και αυτή είναι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Μπορεί να χρηματοδοτούμε το μετρό στη Σόφια της Βουλγαρίας, αλλά αποδέκτε και δικαιούχοι είναι η Βουλγαρία, αλλά είναι και άλλες επιχειρήσεις από άλλες χώρες. Το λέω αυτό για να αποδείξω πόσο κοινά είναι τα συμφέροντά μας. Εμείς ε, ε, στεκόμαστε στο πλάι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέλουμε να ζητήσουμε ένα προπολογισμό φιλόδοξο στο ύψο των περιστάσεων που αναλογεί στην Ευρώπη στο ύψος των προτεραιοτήτων που παρουσίασε η Επιτροπή και η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν εμφανίστηκε ενώπιον σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι νέες προκλήσεις χρειάζονται και νέα μέσα χρηματοδότησης. Πρέπει να ξεπεράσουμε το υφιστάμενο πλαίσιο χρηματοδότησης για να ξεφύγουμε από αυτές τις νοσηρές συζητήσει. Βεβαίως δεν είναι εύκολο αυτό το μέλημα και το εγχείρημα παρόλο που οι εμπειρογνώμονες οι ειδικοί για την ομάδα του ευρώ έχουν συντάξει θαυμάσιες εκθέσεις και ξέρετε οι ομάδες εμπειρογνωμόνων ε, στις, στην Ευρώπη ε, συνέχεια ονομάζονται ευρώ Ποτέ δεν υπόθηκε το αντίθετο. Όμως δεν αντλούμε τα διδάγματα των ε, προτάσεών τους και αυτό ενδεχομένως τους κάνει και κατά τη ήρωες. Σε κάθε περίπτωση οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, αν καταλήξουν σε ένα χαμηλό επίπεδο φιλοδοξιών, εμείς ως Επιτροπή των Περιφερειών θα σταθούμε πλάι σας σε αυτό τον αγώνα για να αλλάξει αυτό το σκηνικό. Η ταχύτητα συχνά βρίσκεται σε αντίθεση με την επίτευξη αποτελεσμάτων και η επίτευξη ισορροπίας είναι κάτι το σημαντικό. Ο κοινός προϋπολογισμός της Ευρώπης είναι γελίος σήμερα για μια ένωση 500 εκατομμυρίων πολιτών. Ζητούμε μεγαλύτερο προϋπολογισμό, μεγαλύτερα περιθώρια επενδύσεων. Και ίσως είναι ένα και από τα θεμελιώδη προβλήματα αυτά, αυτό, όταν μιλούμε για τα οικονομικά μέσα, συχνά Γίνεται λόγος για, το, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα επενδυτικά εργαλεία, τα διάφορα ταμεία και κονδύλια επενδυτικά και όλοι νομίζουν ότι όλα θα λυθούν ως εκθαύματος εάν κάτι μπει σε ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο. Δεν σημαίνει ότι θα αντικαταστήσουμε μία ενίσχυση με δάνειο και θα λυθεί το πρόβλημα. Απλά πάρα πολλά πράγματα περνούν κάπως ε, με μη φανερό τρόπο από το ένα μέρος στο άλλο. Αντί να μιλούμε για ανισχύς, μιλούμε για δάνεια. Σε κάθε περίπτωση ήταν ταμπού όλα αυτά τα θέματα για πολύ καιρό στην ευρωπαϊκή ε, καθεστική ατάξη. Τι εννοώ ο τρόπος υλοποίησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό ήταν ταμπού. Οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας για το έλλειμμα που ε, επιτρέπεται για τα, και τα λοιπά και ο συνδυασμό τους με κανόνες μη λογιστικούς και αντιοικονομικούς ήταν δύσκολος. Το να εμποδίζουμε τα κράτη-μέλη να προχωρούν και να λειτουργούν όπως σε οποιοδήποτε επιχειρηματία σε απόσβαση των δανείων τους, των επενδύσεών τους, είναι κάτι το οποίο ε, δεν λειτουργεί και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πάρει και Νόμπελ οικονομίας. Είναι κάτι που τίθεται υπό αφισβήτηση εδώ και αρκετά χρόνια και νομίζω ότι η λύση στα προβλήματά μας θα προέλθει με ένα ε, νέο τρόπο αναδιάταξης και αναδιαμόρφωσης των τριών βασικών στοιχείων και κεφαλαίων που αποτελούν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αποτελεί προσωπική μου πεποίθηση αυτό. Οι δημόσιες επενδύσεις δεν πρέπει να γίνονται αντιληπτές ως κίνδυνος για την οικονομία μας, αλλά ως αναγκαιότητα για την υποστήριξη της ανάπτυξης. Και τελευταία παρατήρηση, κυρίες και κύριοι, βουλευτές. Για να υλοποιηθούν οι προτεραιότητες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειαζόμαστε απαραίτητα μέσα. Επαρκή μέσα, αλλά και καλές μεθόδους. Αυτό χρειαζόμαστε και πιστεύω ότι οι καλές μέθοδοι βρίσκονται στην πολιτική συνοχή, στη στενή συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης. Και εμείς στην Επιτροπή των Περιφερειών, δεν θα εκπλαγείτε, ε, που μαθαίνετε ότι Συνεχώς απευθυνόμαστε σε όσους, όλους όσοι θέλουν να μας ακούσουν ότι αυτό το πολυεπίπεδο σύστημα, τουλάχιστον τρία επίπεδα, ευρωπαϊκό, εθνικό και επίπεδο ε, τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων με 500.000 κοινότητες, με 300 περιφέρειες στην Ευρώπη, με ε, χιλιάδες ε, δήμους και οτά, είναι ένα σύστημα σημαντικό, είναι μια μέθοδος αυτή, η πολυεπίπεδη, που μας επιτρέπει να διαφοροποιούμε τους ευρωπαϊκούς στόχους αναλόγως με τις ανάγκες που έχουν εκφραστεί στις κατατόπους περιοχές, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, δήμο, πόλη, συνεκία, εκεί όπου μένει ο εκάστοτε Ευρωπαίος πολίτης. Γιατί μπορούμε έτσι να υιοθετούμε εδαφικές προσεγγίσεις, προσέγγιση ανάλογα με την περιοχή και μπορούμε να εμπλέξουμε περισσότερους πολίτες στην ενεργή συμμετοχή για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Έρχομαι τώρα στις προτεραιότητες της κυρίας Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το New Green Deal, η Νέα Πράσινη Συμφωνία. Όλα τα προγράμματα το μεγαλύτερο πρόγραμμα για την οικολογική, μετάβαση δεν είναι το LIFE, ούτε ε, Horizon, ούτε τίποτα άλλο. Είναι το πρόγραμμα της πολιτικής συνοχής, οι επενδύσεις οι τεράστιες στην κυκλική οικονομία, με το 80% των επενδύσεων να επικεντρώνονται στην κοινοτομία και στην κλιματική αλλαγή, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Με την πολιτική συνοχής χτίζεται σιγά σιγά η πράσινη οικονομία του αύριο, η προστασία της βιοπικιλότητας και οι ενεργειακές ζώνες με καινοτόμες μεταφορές. Έχουμε λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, την οποία θα πετύχουμε με την πολιτική συνοχή και έτσι η οικολογική μετάβαση θα συνάδει με την αλληλεγγύη. Η πολιτική συνοχή είναι αυτή που επενδύει πάνω από 110 δις ευρώ σε καινοτόμε δραστηριότητες στο ψηφιακό κόσμο που θα αξιοποιήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι αυτό που επέτρεψε σε 8,9 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες να αποκτήσουν νέα προσόντα και δεξιότητες και επέτρεψε σε 7 εκατομμύρια από αυτούς να βρουν θέση απασχόλησης χάρη σε αυτά. Για να προσαρμοστεί η Ευρώπη στη ψηφιακή εποχή, 20 δις ευρώ επενδύονται στις τεχνολογίες της πληροφορικής, της πληροφορίας και των επικοινωνιών από το 2014 μέχρι και το 2020. Για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η ΟΤΑ που στηρίζονται στην πολιτική συνοχής βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να διευκολύνουν την ένταξη των νέων κατοίκων. Και όταν γίνεται λόγος για μια Ευρώπη πιο ισχυρή στον κόσμο, η πολιτική συνοχής είναι αυτή που θα διαδραματίσει και το πιο σημαντικό ρόλο. Ρόλος ο οποίος αναδεικνύεται στο έγγραφο προβληματισμού για την ε, χειραγώγηση της παγκοσμιοποίησης που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πολιτική συνοχή με τις στρατηγικές έξυπνη εξειδίκευση με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ευρωπαϊκών βιομηχανιών είναι αυτή που αποτελεί και το πιο σημαντικό πόλο στο ευρωπαϊκό τρίγωνο βιομηχανία που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας και θα πρέπει η Ευρώπη να ξανασχοληθεί ουσιαστικά με την έννοια ευρωπαϊκή βιομηχανία, αλλά είναι άλλη συζήτηση αυτή. Και τέλος, όταν γίνεται λόγος για νέα δημοκρατική όθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική συνοχή είναι η πιο επίκαιρη και η πιο σκόπιμη, γιατί είναι η μόνη πολιτική που μπορεί κανείς να υλοποιήσει και αυτό άλλωστε αποτελεί υποχρέωση του κανονισμού είναι η μόνη πολιτική που μπορεί να υλοποιήσει τις αρχές ε, του πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Είναι αναπόδραστο στοιχείο ε, για να παραμείνουν προσκολλημένοι στο ευρωπαϊκό όραμα οι Ευρωπαίοι πολίτες και επιτρέψτε μου να σας πω ότι πρέπει να καταδικάσουμε και να αγωνιστούμε στις πράξεις για να καταπολεμήσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια να γίνει πιο ευέλικτη αυτή η προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. διότι οι εταιρικέ σχέσεις αφορούν όλους. Ίσως είναι στο DNA των κρατών να μην έχουν ε, εμπιστοσύνη στους ΟΤΑ και να θέλουν να έχουν κεντρική διοίκηση στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Ακόμα και ε, τα κράτη που έχουν δημιουργηθεί για να λειτουργούν με όσο το πιο αποκεντρωμένο τρόπο έχουν μια δράνεια, μια τάση να γίνονται όλο και πιο ε, κεντρικά στην ε, προσέγγιση τους. Σε κάθε περίπτωση η πολιτική συνοχή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αποτελεί το ουσιαστικό DNA το συστατικό DNA της Ένωσής μας. Δεν θα μπω στις τεχνικές λεπτομέρειες όλων αυτών τα οποία υπερασπιζόμαστε. Σε κάθε περίπτωση οι θέσεις που υπερασπίζεται η δική μας Επιτροπή συγκλίνουν με τις δικές σας. Είναι εξαιρετική η συνεργασία μας. Γίνονται κοινέ προσπάθειες από τους εισηγητές, από τις πολιτικές ομάδες, από τις γραμματείες για τις νομοθετικές προτάσεις για την πολιτική συνοχής. Και αυτό δείχνει ότι έχουμε συνέπεια και εμείς και εσείς. Ήταν δύσκολο από πλευράς επιμελητίας και από πλευράς οργανωτικής θα έλεγα γιατί έπρεπε και εμείς και εσείς να είμαστε έτοιμοι εγκαίρως, ενώ τα μέλη μας δεν είναι πολιτική πλήρους απασχόληση στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για αυτό. Διατηρούμε τις αρχές της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Είμαστε κατά οποιασδήποτε προσπάθειας να αποδυναμωθεί το άρθρο 6 του κανονισμού περί κοινών εφαρμοστικών διατάξεων, όπως σας υπενθύμησα. Οι συμφωνίες εταιρική σχέσης πρέπει να παραμείνουν υποχρεωτικές για το σύνολο των κρατών μελών. Απορρίπτουμε τις προτάσεις του Συμβουλίου που αφήνουν στα κράτη-μέλη την επιλογή να αξιοποιήσουν ναι ή όχι τα εργαλεία ε, ενσωματωμένης εδαφικότητας. Θεωρούμε ότι αυτά τα εδαφικά εργαλεία είναι εξαιρετικά σημαντικά και πρέπει υποχρεωτικά προς τα εκεί να πηγαίνουν όλα τα, τα κονδύλια για να υλοποιηθούν οι στόχοι της πολιτικής συνοχής και της εδαφικής πολιτικής ατζέντα έτσι όπως έχει ανανεωθεί και αναβαθμιστεί. Ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική δομή που θα πάρουν τα κονδύλια και τα ταμεία στο μέλλον, το 3% πρέπει να στρέφεται προς τη συνοχή των περιφερειών. Το σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά με εσάς για όλα αυτά τα θέματα. Η δική μας Επιτροπή έχει εισηγητές που είναι έτοιμοι να δουλέψουν εντατικά. Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να μας ε, επισκεφθείτε, αλλά και εμείς να συμμετάσχουμε ε, στις συνεδριάσεις της δικής σας Επιτροπής. Έτσι θα αναπτυχθεί έτσι περαιτέρω η συνεργασία μας. Και να ολοκληρώσω θίγοντας ένα θέμα το οποίο συχνά παραμελούμε και το οποίο όμως είναι απαραίτητο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μιλώ για την επικοινωνία. Κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, τον Οκτώβριο, στις ε, εναρκτήριες συνεδριάσεις, οι νέοι αιρετοί ε, είπαν ότι η πολιτική είναι κατά 80% επικοινωνία. Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ απολύτως με αυτά τα ποσοστά, όμως χωρίς επικοινωνία καμία πολιτική δεν μπορεί να επιτύχει. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και ο νέος που το ανέφερε αυτό πράγματι έθεξε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και γι' αυτό στη δική μας Επιτροπή το παίρνουμε πολύ σοβαρά το θέμα αυτό και με, μεγάλες, ε, με μεγάλους συνδέσμους ε, από πλευράς ΟΤΑ ε, έχουμε τη Συμμαχία για την συνοχή όπου συμμετέχουν πάνω από 130 πόλεις και πάνω από 130 περιφέρειες που έχουν υπογράψει και έχουν προσχωρήσει αυτή τη συμμαχία που έχουμε σφυριλατήσει. Μέχρι και η UEFA έχει υπογράψει. Μπορεί κανείς να συζητήσει για το κατά πόσο είναι καλό το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, το επαγγελματικό ή όχι. Εν πάση περιπτώσει ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι για να πούν ότι το, η άθληση έχει σημαντικό ρόλο να διαρροματίσει σε επίπεδο πολιτικής συνοχής. Ετερόκλητη συμμαχία λοιπόν από πάρα πολλούς φορείς ε, κρατικούς και ιδιωτικού συμμαχία για την ε, συνοχή. Έχουμε πάρα πολλούς υπογράφοντες. Επομένως. Κύριε Πρόεδρε, και εσείς, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, υπογράψατε αυτή τη διακήρυξη για τη συμμαχία για τη συνοχή. Θέλω λοιπόν να προτείνω σε όσους ε, μας ακούν αυτή τη στιγμή ε, ε, ότι μπορούν να το κάνουν, μπορούν και εκείνοι να προσχωρήσουν σε αυτή τη συμμαχία μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής των Περιφερειών στο κοινοβούλιο σας. Είναι μια εξαιρετικά ε, σημαντική συμμαχία η οποία έχει ήδη πετύχει πολλά πράγματα. Είχε, ήταν ήδη επιτυχημένη πριν την κατάθεση της πρότασης αυτής από την Επιτροπή και δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες. Όμως, πολλά από τα οποία, πολλά που δεν θα μας έβρισκαν σύμφωνους, δεν υπήρχαν στο αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Δηλαδή ο αρμόδιος επίτροπος έβαλε την μπάλα στη μέση του γηπέδου, στη σέντρα. Δεν μεροληπτήσε, όμως δεν έχουμε ακόμα ε, βάλει αρκετά γκολ. Και θέλω να πω και σε εσά και στους λοιπούς μας εταίρους ότι το αποτέλεσμα θα κρυθεί στο τέλος. Μαραθώνιος είναι. Ξεκινήσαμε πριν από ορισμένα χρόνια. Σιγά σιγά προχωρούμε. Ίσως φτάνουμε στην τελική ευθεία. Και είναι διαφορετικό από τον κανονικό μαραθώνιο, γιατί σαν κανονικό μαραθώνιο ξέρει κανείς πόσο του μένει ακόμα, πόση απόσταση του μένει να διανύσει. Εδώ λοιπόν η γραμμή του τερματισμού σε βάθος χρόνου αλλά και από πλευράς χώρου μπορεί να αλλάξει. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη αθλητική διοργάνωση αυτή και γι' αυτό εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών που θα γιορτάσουμε και την 25η μας επέτειο Λίαν Σύντομος, θέλουμε να κινητοποιήσουμε τους πάντες, θέλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτό τον στόχο. Για αυτό το στόχο. Είναι προς το συμφέρον όλων μας έτσι ώστε στην επόμενη προγραμματική περίοδο να συνεχίσει η πολιτική συνοχής, όπως και στο παρελθόν, να παίζει σημαντικό ρόλο και να βοηθά ιδιαίτερα στην επίτευξη των στόχων μας. Όσοι πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχή είναι μια πολιτική του παρελθόντος, απατώνται, πλανώνται. Είναι μια μέθοδος η πολιτική συνοχή, μια εξαιρετικά καλή μέθοδος, πολυεπίπεδη, για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις τις σημερινές και πρέπει όλοι να εργαστούμε πολύ σκληρά για να πείσουμε όσους δεν έχουν πιστεί ακόμα για την ανάγκη να βρεθεί καλή συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμείς δεν είμαστε στη γραμμή του πυρός, στην πρώτη γραμμή, αλλά ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κινητοποιήσουμε τους υπουργούς και τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και ξέρουμε και πού πρέπει να τους βρούμε. Θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε κίνητρα, να τους πείσουμε. Και αυτή είναι η δουλειά που θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες, μήνες, εβδομάδες. Ελπίζω να μην κρατήσει και χρόνια. Να ολοκληρωθεί αυτό το έργο έτσι ώστε η νέα προγραμματικής περίοδος περίοδο να είναι ακόμα πιο επιτυχημένη από ό,τι στο παρελθόν προ όφελο των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που υπερασπίσατε με τόσο θέρμη, με τόσο θέρμη τη συνοχή. Και θέλω να πατήσω φόρο τιμή στις ε, ακούραστες προσπάθειές σας, ε, κυρίως ε, επί του παρόντος, προκειμένου ε, να συγκεντρώσετε ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη υποστήριξη για τη συνοχή. Και είπατε ότι αυτό είναι ένα έργο που θα πρέπει να επιτελέσουμε τους επόμενες εβδομάδες και μήνες, γιατί διαφορετικά θα είναι πολύ αργά. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα θα έχουν αντίκτυπο στα επόμενα δέκα έτη στη ζωή των Ευρωπαίων και ίσως θα έχουν παντοτινό αντίκτυπο στο μέλλον της πολιτικής συνοχής. Θα ανοίξω τώρα τη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για να ξεκινήσουμε από την κυρία Μαρτίνα Μισελ. Ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Καρχάνης, γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό στο πλαίσιο των εργασιών ε, της ε, Επιτροπής των Περιφερειών, στην οποία συμμετείχα και εγώ για 10 χρόνια. Και κατά συνέπεια εκεί εγώ μεγάλωσα, αν θέλετε, εκεί ορίμασα. Και σε αυτό το πλαίσιο έμαθα και να εκτιμώ βαθύτατα τις εργασίες της Επιτροπής των Περιφερειών. Και εσύ μας ανέφερες τώρα τις νέες ε, προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε και το γεγονός ότι ακριβώς λόγω αυτών των νέων ε, προκλήσεων είναι πιο σημαντικό από ποτέ να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες, να βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους ε, πολίτες ε, και η Επιτροπή των Περιφερειών κάνει ακριβώς, ακριβώς αυτή τη δουλειά, δηλαδή το να προσανατολίζεται να και να εξατομικεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ανάγκες των πολιτών. Και νομίζω εδώ πως θα πρέπει να γίνει κοινή προσπάθεια από τη δική μας πλευρά προκειμένου να αντεταχθούμε στην ε, τάση που υπάρχει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δημιουργούν όλο ένα και πιο κεντρικές δομές. Εμείς λοιπόν από κοινού θα πρέπει να τονίσουμε και να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε τον ρόλο των περιφερειών. Και νομίζω πως θα πρέπει να υπάρξει μια ε, κοινή στρατηγική από δική μας πλευρά έναντι της Επιτροπής και έναντι του Συμβουλίου. Και όποιος με γνωρίζει ε, θα ξέρει ότι το αναφέρω ξανά και ξανά αυτό. Θετώ δηλαδή ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιτρέψουμε στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να συμμετέχουν ενεργά ε, στην λήψη των αποφάσεων και στο σχεδιασμό των διαφορών πρωτοβουλίων. Αυτά τα λέω ε, εισαγωγικά. Ε, τώρα έμαθα ότι θέλεις να συνεχίσεις μόνο μέχρι τα τέλη αυτού του έτους ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, των Περιφερειών. Ε, οπότε από την δική μου πλευρά, αν αυτό ενισχύει, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας, αλλά και προσωπικά ε, για την δουλειά που έχεις κάνει, την αφοσίωση που έχεις δείξει για λογαριασμό της Επιτροπής των Περιφερειών. Και ελπίζω και είμαι βέβαια ότι θα υπάρξει ένας πάξιος διαδοχός ή μία διαδοχός σου δεν θα ήταν ε, άσχημο να είναι διάδοχος, δηλαδή η γυναίκα, έτσι ώστε να συνεχίσουμε αποτελεσματικά τις εργασίες μας ε, και τη συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, όπως αυτή λαμβάνει η χώρα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ, Μαρτίνα, για τους σοσιαλιστές. Ο κύριος Μάρτιν. Κυρία, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για την παρέμβασή σας, αλλά και για την εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μου άρεσε πάρα πολύ η ομιλία σας και κάποιες προσωπικές αξιολογήσεις που κάνατε. Γιατί σίγουρα βρισκόμαστε σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή. Έχουμε την μεταρρύθμιση των ταμείων, τη συζήτηση για το πολιτές πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και έχουμε μεγάλες προκλήσεις. Και αυτή η έκκληση από τους καθαρούς ε, εισφέροντες ε, δεν ε, συνάδει με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα που πρέπει να συμβάλλει ουσιαστικά στην οικοδόμηση του ευρωπαϊκού οράματος. Βέβαια υπάρχει ένας ευρωσκεπτιστικός ε, λόγος που θα έχει σοβαρές ε, συνέπειες ε, και λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συζήτηση αυτή για τις καθαρές εισφορές νομίζω ότι αποτελεί απειλή για τη μελλοντική πολιτική συνοχής. Εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι ότι ε, πέρα από το πώς μπορούμε να δούμε πώς θα βελτιώσουμε ε, τα ταμεία συνεχής, να εξετάσουμε και άλλα ζητήματα που βρίσκονται σε δεύτερο πλάνο. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα δικαιούχο που αντιμετωπίζει σήμερα μεγάλες δυσκολίες σε πάρα πολλές περιφέρειες η υλοποίηση και η εκτέλεση των κονδυλίων ε, λόγω ε, των ε, μεγάλων απαιτήσεων που θέτουν οι κανονισμοί σίγουρα με ανησυχεί. Με ανησυχούν τα εκκρεμή ζητήματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Παίρνοντα χάρη ότι υπάρχει υπερβολική ακαμψία στη θεματική συγκέντρωση, το θέμα της χρηματοδότησης, το θέμα της απλούστευσης των διαδικασιών και θέματα που είναι σημαντικά όπως ε, παραδείγματος χάρη μακροοικονομική αιρεσιμότητα ή ακόμη και σε συγκεκριμένα ζητήματα το γεγονός ότι κάποιες περιφέρειες ε, που χρήζουν κονδύλιων συνοχής θα πρέπει να αιτιολογήσουν ως έλλειμμα ε, τα έσοδα από τα ταμεία Συνοχής. Δηλαδή μπαίνουμε σε έναν φαύλο κύκλο που είναι δύσκολο να αιτιολογήσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, τελικά, αντί να βελτιώνουμε τη ζωή των πολιτών, μπαίνουμε σε έναν ε, κύκλο, φαύλο κύκλο, να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αιτιολογήσουμε τα κονδύλια αυτά. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να μου πείτε τι σκέφτεστε για αυτά τα ζητήματα. Μιλώντας, ε, μιλούμε για τους μικροοικονομικούς κανονισμούς, ε, σαν να πρόκειται για το μαγικό ραβδί και έτσι παρουσιάζονται όντω, αλλά πώς όλοι μαζί, το Κοινοβούλιο, Επιτροπή των Περιφερειών, να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε σε περιοχές όπως στη δική μου στην Καστίγια Λαμάντσα, και στη χώρα μου, την Ισπανία, αλλά και σε πολλές άλλες περιφέρειες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, να μπορέσουμε να προσφέρουμε λύσεις στους πολίτες. Γιατί τελικά μιλάμε για τα συμφέροντα των πολιτών εδώ. Σας ευχαριστώ και πάλι να σας επαναλάβω τα συγχαρητηριά μου. Ευχαριστώ πολύ. Στέφαν Βυζού για το Ρινιού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών. Εγώ είμαι ε, μεταξύ του 60% των νέων ευρωβουλευτών και ξέρω ήδη πόσο σημαντικό είναι το όργανο που προεδρεύεται και μόλις ε, άκουσα ε, ουσιαστικά μια πολύ ευφυή και δυνατή ομίλια από σας και σας ευχαριστώ που τα μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας. Είπατε στην ομιλία σας πόσο σημαντικό είναι για την επικράτεια και για τις απομακρυσμένες περιοχές που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση η σημασία να ξαναβρούμε την ορθή οδό της, των Ευρωπαϊκών Δημοσίων Επενδύσεων. Μιλήσατε για αυτές τις επενδύσεις ως ένα μοχλό ανάπτυξης. Ε, φυσικά ε, δημιουργούν και θέσεις εργασίας ως συνέπεια και το χρειαζόμαστε αυτό τα μάλα. Επίσης, ε, πρέπει να ενθαρρύνουμε τις τοπικές πρωτοβουλίες ε, και είναι πολύ Πολύ συχνά προσκρούν ε, σε δυσκολίες στην πολυπλοκότητα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Διοίκησης. Θέλω να σας ρωτήσω αν η οδή απλούστευσης, γιατί η απλούστευση δεν αποκλεί τον έλεγχο, αλλά ο περιβολικός έλεγχος σκοτώνει τις πρωτοβουλίες και θέλω λοιπόν βάσει της εμπειρίας σας να σας θέσω αυτή την ερώτηση γιατί πολλές φορές αναφερθήκατε στην ανάγκη να έχουμε τις καλές μεθόδους. Ποια είναι η ορθή μέθοδος κατά την άποψή σας για να πετύχουμε την επλούστευση της δέσμευσης της Ευρώπης έτσι ώστε να εξυπηρετήσει, να υπηρετεί τις περιφέρειες. Ευχαριστώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Από τους Πρασίνους ο κύριος Αλφόνση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και για τη δική σας ε, παρέμβαση διαπιστώσαμε ότι συγκλίνουν ε, τα μέλη απόψεις μας. σε σχέση με τα όσα μας απασχολούν. Είναι κάτι και εκτιμένο, όμως είναι σημαντικό νομίζω να το τονίζουμε όπως γίνεται και σήμερα. Πέρα από αυτή τη σύγκληση στους στόχους, μήπως θα μπορούσαμε να δούμε τι σύγκληση μπορούμε να έχουμε και στις διαδικασίες. Δηλαδή να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Στη έγγραφα που έχω λάβει της Επιτροπής των Περιφερειών υπάρχει μια πρόταση που διατυπώσατε που τράβηξε την προσοχή μου. Δεδομένου του γεγονό ότι η κυρία Φοντελάιεν αναφέρθηκε στην δυνατότητα να υπάρχει ένα τριπλό Εράσμους από την Ισομική Σκοπιά. Η Επιτροπή των Περιφερειών ε, θα προτείνει ένα Εράσμους ε, ε, δαφικό που να μπορεί να υλοποιηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή είναι μια πρόταση με την οποία συμφωνούμε και θα ήθελα την άποψή σας με το πώς μπορούμε από κοινού να την προωθήσουμε προκειμένου να υλοποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας δώσω το λόγο, κύριε Πρόεδρε, για να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και για τις ερωτήσεις σας που επιβεβαιώνουν καταρχήν το θέμα της σύγκλησης. Δεν συμφωνούμε πάντα με όλους όμως ε, υπάρχουν θεμελιώδη δακευμένα όπου επιβάλλεται η σύγκληση. Και η σύγκληση αυτή ήδη τη βιώνουμε πέρα από τα όρια, τα σύνορα των διαφορών πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή των Περιφερειών. Γιατί εδώ έχουμε κάτι κοινό σε όλους. Όταν ε, έχεις εκλεγεί σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να είσαι ρεαλιστής υποχρεούσε να είσαι ρεαλιστής. Και συχνά καλείσαι να περάσεις ε, κάποιους θεωρητικούς ε, ενδιασμούς ε, και να συνεργαθείς με τους συναδέλφους. Εγώ τουλάχιστον ε, τα έτη, τα τελευταία έτη που είμαι μέλος Επιτροπής των Περιφερειών από την αρχή Τη χιλιετία μπορώ να σας πω, πάντοτε αυτό που με εξέπλητε εκεί ήταν η δυνατότητα να βρίσκουμε συνένεση για ιδιαίτερα επίμαχα θέματα σε ό,τι αφορά τη γενική πολιτική. Αυτό το βιώσαμε σε αυτό το κεντρικό ζήτημα και στο κείμενο που έχουμε προετοιμάσει αναφέρθηκε. μιλώ για το θέμα της ε, διαχείρισης της δίκησης ε, σε μια περιφέρεια. Μπορεί να γίνει και υπό τη μορφή ενός ε, εργαστηρίου να υπάρχει ένα συνδυασμός εφιούς πολιτικής μιας εφιούς πολιτικής χρήσης ενός χρηματοοικονομικού εργαλείου που να έχει αποτελέσματα μόχλευσης αλλά και επιστροφής των μέσων στη συνέχεια και ταυτόχρονα ρεαλιστικής, ευέλικτης υλοποίησης κριτηρίων του Συμφώνου σταθερότητα. Ο συνδυασμός μεταξύ αυτών των τριών στοιχείων είναι ουσιαστικός και είναι ένα πολύ μεγάλο στοιχείο που συμβάλλει στην επιτυχία. Και φυσικά χρειάζονται προσπάθειες όλων. Μερικές φορές κάποιοι είναι δύσκολο να πιστούν. Στα γερμανικά λέμε ότι θέλουμε πάντοτε να είμαστε σε θετικά νούμερα. Εκεί πρέπει να έχουμε κάποια εξέλιξη, αλλά πρέπει να έχουμε και εξέλιξη ό,τι αφορά το επίπεδο των διαχειριστών. Θα πρέπει να καινοτομούμε, να είμαστε δημιουργικοί. Και Παραδείγματο χάρη, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπάρχει εξαιρετική τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά το middle management και θα ήμασταν πολύ ευτυχεί. αν ε, μας το ζητούσαν περισσότερες φορές ε, για να συμμετέχουμε από την αρχή στην ε, πραγματική οικοδόμηση των προγραμμάτων. Νομίζω ότι έχουμε πολύ σημαντική δουλειά να κάνουμε εκεί, αλλά σίγουρα, όπως ε, κάποιοι ήταν, μπορούμε να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία πλουστεύοντας τους κανόνες. Κάθε φορά, σε κάθε νέα περίοδο χρηματοδότησης, υποσχόμαστε την απλούστευση των κανόνων. Το αποτέλεσμα τελικά είναι πάντα το ανάποδο. Την πολυπλοκότητα ακόμη και στην εδαφική συνοχή, που γνωρίζω λεπτομερέστερα, πιστεύω ότι ε, τα σημερινά κείμενα μπορούν να απλουστεύσουν κάποια πράγματα. Αυτό όμως δεν είναι μόνο πρόκληση για τους Ευρωπαίους νομοθέτες, αλλά και για τους ανθρώπους που λειτουργούν επί τόπου. Εγώ έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη διασυνοριακή ε, συνεργασία και ήμουν πρόεδρος του οργανισμού για τις συνοριακές περιοχές. Βλέπαμε ότι είναι δύσκολο να υλοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες και για να γίνει αυτό θα έπρεπε να βάλουν δύο διαφορετικές αιτιολογίες οι αρμόδιοι. Αυτό είναι κάπως ιδιαίτερο πάντοτε. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Η μεγάλη συζήτηση είναι αυτή της αλληλεγγύης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη αυτή. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η λέξη. Αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε και μια αγαθή προσέγγιση. Συχνά η αλληλεγγύη αντιμετωπίζεται απλουστευτικά, ότι είναι οι πιο πλούσιοι, που δεν είναι και τόσο χαρούμενοι να δίνουν χρήματα στους πιο φτωχούς. Υπάρχει και αυτή η διάσταση, όμως η πραγματική αλληλεγγύη είναι το κοινό συμφέρον. Αν θέλουμε σε αυτή τη μικρή πυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη αν θέλετε, ο Νέος είναι πιο μικρή, να πάμε πιο πέρα από τα εθνικά σύνορα, αν θέλουμε να πετύχουμε σήμερα και αύριο παγκοσμίω, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο συνεκτικοί. Η συνοχή είναι κάτι εντελώς απαραίτητο και αυτή η συνοχή θα πρέπει να συνεισφέρει έτσι ώστε να έχουμε μια παρόμοια κατάσταση σε όλη την Ήπειρο. Και είναι πραγματική δουλειά που πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει πάντοτε να το αναφέρουμε και θα πρέπει να το μεταφέρουμε και στην πραγματικότητα, γιατί ωραία τα λέμε στα λόγια, αλλά όταν πρέπει να περάσουμε στις πράξεις δυσκολεύουν τα πράγματα. Για μένα το Brexit ήταν μια τεράστια απογοήτευση, όπως για όλους. Παρ' όλα αυτά έμαθα δύο πράγματα. Εδώ και κάποιο καιρό θαυμάζω βαθιά Ε, τον πρόεδρο του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Και το λειτουργήμά του χθε το βράδυ, μάλιστα, συγκινήθηκα όταν στο Westminster διόρισαν τον ε, καινούριο. Ε, μπορούμε να δούμε ότι εκεί μπορούν να συμφιλειωθούν κάποιες δυσκολίες της δημοκρατίας. Όμως κάτι άλλο που κόπως με παρηγορεί μέσα σε όλη αυτή την υπογοήτευση που νομίζω και εσείς συμμερίζεστε είδα και βίωσα με πάσα λεπτομέρεια πως ε, ο Πρωθυπουργό της ε, Βρετανίας χειρίστηκε όλο αυτό το θέμα του δημοψηφίσματος. Αποτελεί ένα μεγάλο λάθος, σοβαρότατο λάθος. Όμως αυτό που ζήσαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό που θα συνεχίσουμε να βιώνουμε αποδεικνύει το εξή. Πέρα των ε, κακών που μπορούμε να αποδώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι τόσο εύκολο κανείς να την εγκαταλείψει. Και όταν την εγκαταλείπει, συνειδητοποιούμε ότι όλοι είμαστε χαμένοι. Και νομίζω, και τουλάχιστον το ελπίζω, ότι αυτό θα έχει μία επιρροή στους υπόλοιπους 27 και ίσως ε, και στις άλλες χώρες ε, που θα προσχωρήσουν σε κάποιο καιρό. Εμείς ε, λυπηθήκαμε πάρα πολύ σε Επιτροπή των Περιφερειών όταν ακούσαμε την απόφαση που αφορούσε την προσχώρηση της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Μάλιστα εγώ λίγες μέρες πριν είχα συναντήσει ε, Πολλού ε, υπεύθυνου στον κροτικό μηχανισμό της Βορειάς Μακεδονίας και πολλοί στεναχωρήθηκαν. Νομίζω ότι εδώ κάναμε ένα σοβαρό λάθος. Γιατί μιλάμε για μια πολύ στρατηγική περιοχή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αλλά αυτό είναι ένα επιμέρους ε, σχόλιο, ένα παράπλευρο σχόλιο. Δεν συσχετίζεται με την πολιτική συνοχή, αλλά πραγματικά άπτεται τη μελλοντική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η επενδυτική ικανότητα των συλλογικοτήτων των περιφερειών. Ε, ουσιαστικά αυτή η ικανότητα που φτάνει στο 60% του συνόλου είναι πολύ σημαντική. Είναι θεμελιώδης. Αν ε, θέλουμε μεγαλύτερη προσχώρηση στο ευρωπαϊκό ιδεώδες, θα πρέπει η Ευρώπη να συνεισφέρει σε ευφυείς επενδύσεις. Αυτό συζητήθηκε και στο επίπεδο στον οποίο όλοι μιλάνε για smart investment. Δεν έχω ακούσει ποτέ να μιλούν για χαζές επενδύσεις. Αλλά εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτές οι επενδυτικές ικανότητες να ενεργοποιηθούν εκ νέου. Φυσικά όταν θα έχουμε και ένα εύρωστο προπολογισμό. Δεν θα πρέπει να κάνουμε ό,τι να είναι, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό για την τοπική αυτοδιοίκηση όπως είναι πολύ σημαντικό και η τοπική αυτοδιοίκηση να μπορεί να διαχειριστεί τις υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος. Γιατί είναι πραγματικά η ουσία, εκεί έγκυται η ουσία αυτού που γίνεται επί τόπου. Και ακόμη και στις πλούσιες, στις πολύ πλούσιες περιοχές ε, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που δεν ε, μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση, μια αξιοπρεπή κατοικία. Νομίζω ότι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό σε όλα τα επίπεδα εξουσία λοιπόν να το προβλέψουμε. Και για να έρθω και σε μία άλλη πρόταση. Αυτό το τριπλό εράσμο είναι κάτι πολύ καλό. Σε την ε, Κυριακή συμμετείχα σε μια εκδήλωση ε, στη Γερμανία, κοντά στο Βερολίνο και έγινε κάτι πολύ συγκινητικό. Μετά από την ομιλία μου με πλησίασε ένα ζευγάρι και είχαν και ένα μικρό παιδάκι μηνών. Ήταν ένα παιδί Εράσμους. Αυτό πραγματικά με συγκίνησε. Και μου διηγήθηκαν όλοι τους ε, την εμπειρία και πολλοί άνθρωποι μιλούν για τις εμπειρίες τους, ε, πόσο ανοίγει το μυαλό τους, το πνεύμα τους όταν συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα Εράσμους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τριπλασιάσουμε τις ε, προσπάθειες, να διευρύνουμε επίσης ε, τις προσπάθειες για να καλυφθούν και άλλοι πέραν των πανεπιστημίων. Και Επίσης, αν θα μπορούσαμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτή την ιδέα που γεννήθηκε στην Επιτροπή των Περιφερειών, αυτό το Εράσμους των ε, υπευθύνων τη τοπική αυτοδιοίκηση και των ανθρώπων που εργάζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση να υλοποιηθεί έτσι ώστε να μάθουν και τι γίνεται κι αλλού. Και αυτό θα ήταν πολύ καλό. Νομίζω ότι τον οργανώνουμε αυτέ τι ανταλλαγέ. Δεν είναι ένα μεταμφιασμένο τρόπο να εργανώνει κανεί τι διακοπέ του. Αν γίνεται ορθά, πρόκειται για άνοιγμα του μυαλού. Και δεν μπορεί αυτό να αξιολογηθεί με όρους χρήματος, αλλά είναι κάτι ουσιαστικό αν θέλουμε να εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταίο μου σχόλιο. Θέλω να ευχαριστήσω όσους ε, μας συνέχαραν για το έργο μας. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν ε, απλό να κάνει ε, καλή, δουλειά στην Επιτροπή των Περιφερειών, γιατί έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, είναι πολύ καλό το κλίμα. Και κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας ε, η οποία έχει, ε, δεν συμπίπτει κατά 8 μήνες με την θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από την 1η ε, Νοεμβρίου έχουμε μια νέα επιτροπή που θα μπορούσε να μας διαβάσει όλες τις εμπειρίες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή είναι κάπως διαφορετικό το χρονοδιάγραμμα. Παρ' όλα αυτά, θα γιορτάσουμε την επέτειό μας 4 και 5 Δεκεμβρίου για τα 25 έτη της ύπαρξής μας. Λοιπόν, το θέμα της κοινωνίας είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά ε, ζούμε κατά κάποιο τρόπο, ε, βιώνουμε τις διαδικασίες παράλληλα με τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμείς έχουμε αυτή την αλλαγή του Πρόεδρου κάθε μισή έτη και φυσικά εγώ συμμερίζομαι την ιδέα αυτή, αν και αυτό σημαίνει ότι δεν θα είμαι πλέον ε, πρόεδρος από την 1η Φεβρουαρίου του 2020, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την εναλλαγή. Όμως, είναι σημαντικό και το εξή. Να λέμε, δεν θα έχουμε προεδρίες που απλώς θα ακολουθεί μία την άλλη, θα έχουμε μία ομάδα. Δηλαδή, ο πρώτος αντιπρόεδρος ε, ε, και ο πρόεδρος που θα που αλλάζει στη μέση τη θητεία. Συμφώνησαν με το σύνολο των πολιτικών ομάδων και τη διάσκεψη των Προέδρων να σχηματίσουν μια ομάδα και να έχουν ένα πενταετή προγραμματισμό. Γίνεται επιμερισμός των ευθυνών και αυτό έχει αποτελέσει απόλυτη επιτυχία. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που ο συνάδελφο Μαρκολέ από τη Φιλανδία ε, ξεκίνησε αυτή την πρακτική που μπορούσα εγώ να συνεχίσω και εδώ νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα σημαντικό έργο. Η Επιτροπή των Περιφερειών, στα 25 χρόνια που υπάρχει, ξεκίνησε από τις μεγάλες ιδέες ε, μέχρι τις ε, ψευδεστήσεις, ε, απογοητεύτηκε, είχαμε και κατάληψη αν θέλετε και μετά βρήκαμε το δρόμο μας όμως το σημαντικό είναι και ενίοτε τελείως τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη ελληνική πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το είπα, ότι εδώ δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε τον οποιοδήποτε. Είμαστε εδώ για να σα υπενθυμίζουμε συνεχώς όταν μας ρωτάτε, αλλά και όταν δεν μας ρωτάτε, ποιο είναι ο αντίκτυπος της Ευρώπης σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκηση. Και εδώ όλοι εποφελούνται γιατί ουσιαστικά και εκεί έγκυται η Ευρώπη, πέρα από την ε, ωραία πόλη του Στρασβούργου, των Βρυξελών του Λουξεμβούργου, αλλά η Ευρώπη ουσιαστικά που βρίσκεται εκεί που ζουν οι άνθρωποι, στα χωριά, στις πόλεις και στις περιφέρειες. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο στα πολύ σημαντικά λόγια σας αποτελούν έμπνευση για μας να συνεχίσουμε να προβληματιζόμαστε και εύχομαι κάθε μία από τις προτάσεις σας να αναλυθεί από τους συναδέλφους, γιατί είπατε πολύ σημαντικά πράγματα για το μέλλον της Ευρώπης. Όμως, θέσατε και το θέμα της συνοχής σε μία προοπτική, σε ένα όραμα και ακριβώς αυτό μας χρειάζεται. Έτσι λοιπόν, εξ ονόματος όλων των συναδέλφων, σας ευχαριστώ εκ νέου και εκ νέου θέλω να σας πω πόσο πολύ εκτιμούμε και έχουμε εκτιμήσει τη δική σας δράση ως Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών. Σας ευχαριστούμε ένθερμα από την πλευρά της δικής, της δικής μας Επιτροπής. Και Επίσης, ακούσαμε και τη διαθεσιμότητα της Επιτροπής των Περιφερειών να δοθεί συνέχεια στα αιτήματά μας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Δύο λόγια θέλω να σας πω. Επιστρέφω στην Επιτροπή Περιφερειών μέσα από την Πασαρέλα που ενώνει τα δύο κτίρια. Εδώ και πέντε χρόνια κάθε φορά που παίρνω αυτό το δρόμο χάναμε και γι' αυτό συνοδεύομαι από κάποιον που μου το δείχνει. Και το έχω φιλοσοφήσει το θέμα. Εάν θέλει κανείς να καταλάβει τη πολυπλοκότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκεί να ακολουθήσει την παρσαρέλα που ενώνει Ευρωπαϊκή η Επιτροπή των Περιφερειών και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, να, τον, να ακολουθήσετε κι εσείς αυτή τη διαδρομή, να δείτε αν θα χαθείτε όπως εγώ. Σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ. Νομίζω ότι ήταν μια συνεδρίαση η οποία είναι πολύ καλή και πρέπει να υπογράψετε τη Συμμαχία για τη Συνοχή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, το έχω κάνει. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που να αγνοούν αυτή την συμμαχία για τη συνοχή. Όσο περισσότεροι το ξέρουν, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι. Περνούμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων για την απαλλαγή 2018, για τη χρήση 2018. Τελευταίο στάδιο του κύκλου ζωής του προϋπολογισμού είναι η διαδικασία της απαλλαγής, το ξέρετε για δεδομένη οικονομική χρήση, δημοσιονομική χρήση. Ε, η Επιτροπή η Αρμόδια Δημοσιονομικού Ελέγχου ετοιμάζει τη διαδικασία απαλλαγής και έχει να κάνει με όλα τα θεσμικά όργανα και οι υπηρεσίες που λαμβάνουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να χορηγήσουμε την απαλλαγή, να την μεταθέσουμε χρονικά ή να αρνηθούμε την απαλλαγή. Η Επιτροπή Ρέτζη θα θυμάστε ότι αποφάσισε να εκπονήσει μια γνωμοδότηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Επιτροπής για το τμήμα 3 του προϋπολογισμού που είναι το 95% του συνόλου. Η αρμόδια εισηγήτρια θα μας παρουσιάσει τους πρώτους προβληματισμούς για το θέμα αυτό. Θα έχουμε τη χαρά να την ακούσουμε για το σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή μας στις 4 και 5 Δεκεμβρίου. Σας δίνω το λόγο, παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω ε, κάθε χρόνο, η δική μας Επιτροπή καλείται να γνωμοδοτήσει επί της ε, απαλλαγή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ε, της, του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε θα ήθελα σήμερα να σας παρουσιάσω συντομία τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στη γνωμοδότησή μας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της πολιτικής συνοχής. Η δαπάνη σε αυτούς τους τομείς, δηλαδή για ζητήματα οικονομικής κοινωνικής ε, ε, συνοχής, δηλαδή ε, το τίτλος 1β, έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι καμία από τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα αποκλειστεί από την ανάπτυξη, έτσι ώστε να κινηθούμε σε μια ταχεία μείωση των διαφορών ε, που υπάρχουν ε, μεταξύ των διαφορετικών περιοχών. Και αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσω των αναπτυξιακών τομείων, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το 2018 το ελεκτικό συνέδριο έλεγξε 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ ως δαπάνες ε, οι οποίες δαπανήθηκαν σε αυτό το τομέα. Δηλαδή τρεις φορές υψηλότερο αυτό το ποσό σε, σχέση, σε σύγκριση με αυτό που ελέγχθηκε το 2017. Επιτρέψτε μου να τονίσω μια σημαντική πτυχή, η οποία ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη συζήτηση και η οποία παρόλα αυτά θα πρέπει να αναφερθεί, δηλαδή το επίπεδο σφάλματος. Το ελεγκτικό λοιπόν συνεδρίο σε ό,τι αφορά αυτό τον τίτλο, τον 1β, ε, υπολόγισε το επίπεδο του σφάλματος στο, στην τάξη, του 5%. Δηλαδή, αύξηση στο επίπεδο του σφάλματος ε, σε σχέση με το 2017 που ήταν το 3% και μια ε, ελαφριά αύξηση σε σχέση με το 2016 που ήταν 4,8%. Δηλαδή αυτή η θετική τάση ε, έχει ουσιαστικά μειωθεί. Τώρα, εξετάζοντας αυτόν τον ε, προπολογισμό, θα πρέπει να δούμε πως ο, ο που εστιάζει στην ε, πολιτική, οικονομική και εδαφική συνοχή παρουσιάζει και το υψηλότερο επίπεδο σφάλματο. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ένα επίπεδο σφάλματος από μόνο του δεν καταδεικνύει ότι υπάρχει σφάλμα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το στατιστικό μέγεθο, το υπολογισμόμενο ποσοστό, το οποίο καταβάλλεται από το προπολογισμό προ του δικαιούχου χωρί να υπάρχει πλήρης ε, συμμόρφωση με τα συγκεκριμένα κριτήρια. Εμείς όμως ε, ως αρμόδια επιτροπή σε ό,τι αφορά την απαλλαγή, προφανώς θα πρέπει να εξετάσουμε το γιατί ακριβώς έχει προκύψει αυτό το ε, επίπεδο σφάλματος. Με βάση λοιπόν τη σχετική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού σε σχέση πάντοτε με το δημοσιονομικό έτος του 2018, η, τα σφάλματα που έγιναν σε ό,τι αφορά τις ε, περικοπές είναι τα 44% σε ό,τι αφορά τα μη επιλέξιμα project, 14% σε ό,τι αφορά την παραβίαση των ε, κανόνων της εσωτερικής αγοράς και 11% σε ό,τι αφορά ή λόγω της απουσίας των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στο επίπεδο της απορρόφησης ε, των ε, κονδυλίων που αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα και επί του οποίου θα έπρεπε να εστιάσουμε στη γνωμοδότησή μα σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού. Ο εν λόγω λοιπόν δείκτη τη απορρόφηση εξετάζει τον λόγο μεταξύ των κόντιλιο που έχουν καταβληθεί σε έναν δικαιούχο ή σε μια ομάδα δικαιούχων με το συνολικό με βάση την σχετική έκθεση του Ελεκτικού Συναδρίου για το 2018 πάντοτε και την εκτέλεση του προπολογισμού, διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιε βελτιώσει προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο τη απορρόφηση ε, των ε, κονδυλίων των Ευρωπαϊκών Επενδυτικών και Διαθετικών Ταμείων. Έω τα τέλη του 2018, μόνο το 27,3% των συνολικών ε, κονδυλίων σε ό,τι αφορά το σύνολο του πολιτικού διευθυντικού πλαισίου είχαν καταβληθεί, είχαν εκταμιευθεί προ τα κράτη-μέλη. Και το συγκεκριμένο ποσοστό είναι χαμηλότερο από αυτό του 2011 δηλαδή το αντίστοιχο σε σειρά έτος του προηγούμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου του 2007 έως 2013. Μόνο σε ορισμένα δηλαδή κράτη-μέλη αυξάνεται η απορρόφηση των ε, κονδυλίων, ε, των διαθωτικών και επενδυτικών ταμείων σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν ε, το ζήτημα αυτό της απορρόφησης των κοντιλιών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά γιατί αυτή η επιβράδυνση του ποσοστού του, της απορρόφησης σημαίνει ότι προς το τέλος του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου να έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση της ε, απορρόφησης και αυτό ε, θα σήμαινε ότι αυτό θα ήταν αυτό σκοπό κατά κάποιο τρόπο, χωρί ε, να προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την τήρηση των ε, αντίστοιχων ε, ε, στόχων. Οπότε λοιπόν, μια καλή συνεργασία ανάμεσα στι Εθνικέ Αρχέ και την Επιτροπή, καθώ και η σωστή επιβολή του κανονιστικού νομοθετικού πλαισίου, μπορεί να μα βοηθήσει να αποφύγουμε το να συμβεί κάτι αντίστοιχο στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάτι ακόμα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στη γνωμοδότησή μας είναι ο ρόλος των εθνικών ελεγκτικών αρχών και ο ρόλος δηλαδή που παίζουν και αποφασιστική σημασία ρόλο σε ό,τι αφορά αυτά τα κονδύλια. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το δημοσιονομικό έτος του 2018, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο υπογράμμισε ότι υπάρχουν αδυναμίες οι οποίε σχετίζονται κυρίω με τι μεθόδου εργασία που ακολουθούν ορισμένε από αυτέ τι εθνικέ ελεγκτικές αρχέ, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τι μεθόδου δεχματοληψίας αλλά και την τεκμηρίωση των διαφόρων βημάτων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο τη διαδικασία αξιολόγηση. Παρά λοιπόν το γεγονό ότι σημειώνονται διάφορε βέλτιστε πρακτικέ, χρειάζονται ακόμα περαιτέρω βελτιώσει. Τέλο, θα ήθελα να αναφέρω κάτι που ήδη έχω αναφέρει στο πλαίσιο της ε, διαδικασίας απαλλαγής του προπολογισμού του 2017 και είναι η ανάγκη του να υπάρχει ένα σύστημα ε, μέτρησης επιδόσεων το οποίο θα λειτουργεί εύρυθμα και ομαλά. Εάν θέλουμε δηλαδή πραγματικά να είμαστε σε θέση να μετρήσουμε τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να έχουμε δείκτες οι οποίοι θα μας παρέχουν τις κατάλληλες ε, πληροφορίες και θα βασίζονται σε αξιόπιστα και υψηλής σε δεδομένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και αναμένω με ενδιαφέρον τις ε, τοποθετήσεις των σχεδόν εισηγητών και των ε, συναδέλφων προκειμένου να καταρτήσουμε ένα κείμενο γνωμοδότηση το οποίο θα αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητε τη Επιτροπής μας. Merci beaucoup pour ces premières réflexions qui sont déjà... Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πρώτες ε, σκέψεις που προκρίνουν ότι θα είναι καλό το σχέδιο της γνωμοδότηση Να δώσουμε το λόγο στους κοιόδης εισηγητές, ο κύριος Πυρνά Γετορνιού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την πολύ συζήτηση που κάνουμε, για αυτή την γνωμοδότηση και αναμένω με ενδιαφέρον τη συνεργασία που θα έχουμε με τους συναδέλφους. Στις ε, παρατηρήσεις ε, που έκανε πρόσωπος του ε, ελεγκτικού συνεδρίου αναφέρθηκε ακριβώς αυτό το επίπεδο σφάλματος και συμφωνώ με αυτό που είπε τώρα ε, ε, εισηγήτρια ότι δηλαδή το επίπεδο σφάλματο δεν σημαίνει αυτομάτω και σφάλμα. Αυτό δηλαδή οφείλεται ε, συχνά στο γεγονό οτι ότι κάποια κράτη-μέλη προσπαθούν να προσθέσουν κάποια στοιχεία στον κανονισμό. Οπότε εμεί, από την πλευρά τη Επιτροπή Περιφερειακής ανάπτυξη, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τον πολιτικό αντίκτυπο που θα έχει η δική μα τοποθέτηση. Για παράδειγμα, είδα από την πλευρά του ελεκτικού συνεδρίου το παράδειγμα σε ό,τι αφορά τι ε, κάτω χώρε και το πώ δηλαδή εκείνε προσέθεσαν ακριβώ ε, στοιχεία στον κανονισμό δημιουργώντα ε, ιδιαίτερη σύγχυση σε σχέση με του δικαιούχου. Συχνά λοιπόν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι των κρατών μελών κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα σφάλματα που οι ίδιοι έχουν κάνει. Και συχνά βέβαια δεν είναι και ξεκάθαρο το τι συμβαίνει ακριβώ, αν δηλαδή ένα σφάλμα έχει προκύψει λόγω ακριβώ του κανονιστικού ευρωπαϊκού πλαισίου ή λόγω σφαλμάτων για παράδειγμα που των εθνικών κοινοβουλίων ή των εθνικών αρχών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια διαφοροποίησης των, των ε, πραγμάτων, δηλαδή του να υπάρχουν, να διαφοροποιούνται, να είναι ξεχωριστά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτή την κατάσταση όπου θα μας κατηγορούν δηλαδή στο μέλλον για σφάλματα και ε, βήματα που έχουν κάνει οι εθνικές κυβερνήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ε, συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο από τι άλλε πολιτικέ ομάδε Γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιοι θα είναι οι σκιώδει συζητητέ. Παρακαλώ, συνάδελφο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε τον προπολογισμό του 2018 Τώρα βρισκόμαστε στη μέση της περίοδου 2014-2020 και θέλω να πω το εξή. Ακούσαμε ότι καμία περιφέρεια δεν πρέπει να ξεχαστεί. Το 2016 Κάποιες χώρες άλλαξαν ε, το διοικητικό του σύστημα, συμπεριλαμβανομένης και της Λιθουανίας. Όμως, σε ό,τι αφορά την προγραμματική περίοδο 2021-2027, μας ε, λένε ότι τα στατιστικά στοιχεία δεν έχουν συλλεχθεί ακόμα επαρκώς. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το διοικητικό σύστημα στα κρατη και τα στατιστικά στοιχεία, γιατί αυτά θα έχουν αντίκτυπο σε δημοσιονομικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τώρα το επίπεδο σφάλματος. Διαπιστώνουμε ότι αυξάνεται το επίπεδο σφάλματος σε κάποιους τομείς. Ακόμη και αν το γενικό ποσοστό σφάλματος ε, τίνει να μειώνεται. Το γενικό επίπεδο σφάλματος ε, τίνει να μειώνεται. Ίσως ε, θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι περιπτώσει απάτη. Γιατί σε ορισμένε περιπτώσει όντω πρόκειται για απάτη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η πτυχή αυτή. Σε ό,τι αφορά τα όρια σε εθνικό επίπεδο, έχουμε πει ότι μια υπερβολική ευελιξία, μια μεγάλη ευελιξία οδηγεί στα κράτη-μέλη να βάζουν διάφορα όρια και περιορισμούς και να αυξάνουν το διοικητικό άχθος. Γι' αυτό το λόγο η αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων καθυστερεί για πολλά έτη και κατόπιν υποχρεούμαστε να υλοποιούμε τα προγράμματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στο τέλος δηλαδή της διαδικασίας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υλοποιήσουμε έναν ελεγκτικό μηχανισμό για να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. εγκρίνουμε τον ΙΣΙΝΤΡΙΑ 3 και ίσως εξαιτία αυτού υπάρχει έλλειψη ανάληψης ευθυνών. Ο μηχανισμός ΙΣΙΝΤΡΙΑ 3 θα έπρεπε να εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Και αν τα κρατημέλη δεν είναι σε ετοιμότητα να το πράξουν αυτό, ίσως δεν θα έπρεπε να εφαρμόζουμε τον νησί 3. πιστεύω ότι σε εθνικό επίπεδο τα πιο σημαντικά πράγματα συμβαίνουν σε επίπεδο κυβέρνησης. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να εμπλέξουμε περισσότερο και το κοινοβούλιο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τα κοινοβούλια και μάλιστα τα περιφερειακά κοινοβούλια. Γιατί τα κοινοβούλια είναι παρατηρητές αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαν όμως να διαδραματίσουν ένα σημαντικότερο ρόλο, κυρίως όταν η κεντρική κυβέρνηση δεν κάνει τα πράγματα όπως πρέπει ή ξεχνά κάποια πράγματα. Νομίζω ότι θα μπορούσε η συμμετοχή των κυρβουλίων να διευκολύνει τη διαδικασία και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από τις πολιτικές ομάδες ε, να μας στείλουν ε, τα ονόματα των διάφορων σκιών εισηγητών, έτσι ώστε η συνάδελφος ε, να μπορέσει να υλοποιήσει το έργο της με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και να παρουσιαστεί η έκθεση στην επόμενη συνεδρίαση 4 και 5 Δεκεμβρίου. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώνουμε εδώ τη συνεδρίασή μας. Να σας πω ότι η συνεδρίαση των συντονιστών έλαβε χώρα χθες. Έχουμε στείλει και το έγγραφο των αποφάσεων και αν δεν υπάρχει αντίρρηση από εσά, θεωρούμε ότι εγκρίνονται οι αποφάσεις αυτές. Θα τα ξαναπούμε στις 4 Δεκεμβρίου, στις 2 και μισή για μια πρώτη συνεδρίαση και στις 5 Δεκεμβρίου στις 9 το πρωί για τη συνέχεια της συνεδριασής μας. Καλή υπόλοιπη εβδομάδα και στο Πανεδίν.